Κυρίε και κύριοι, σα καλωσορίζω όλου θερμά. Σήμερα έχουμε να εξετάσουμε ένα πραγματικά σημαντικό θέμα και δυστυχώ ε, άλλαξε λιγάκι το χρονοδιάγραμμα. Δεν το θέλαμε, αλλά δεν γινόταν αλλιώ. Υπάρχουν γεγονότα στον κόσμο ναι. που μερικέ φορέ μα αναγκάζουν να αντιδράσουμε. Γι' αυτό στι 5.30 είπαμε να έρθει εδώ ο κύριο Ότιγκερ, που σημαίνει ότι στις 5.30 πρέπει να έχουμε τελειώσει με την ακρόαση. Ε, θα είμαστε όλοι φιντολοί στα λόγια. Εγώ δίνω το καλό παράδειγμα. Λέω καλωσορίστε και τέλος. Και δίνω το λόγο στον κύριο Σούζαν Βάκλα, ο οποίος θα κάνει ίσως κάποιες ε, παρατηρήσεις, γιατί είναι ο εισηγητής για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Η σειρά σας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε και τη δυνατότητα να μιλήσω. Φρονώ όμως ότι ο χρόνος ε, μας είναι πάρα πολύ περιορισμένος, ε, διότι έγιναν αρκετές αλλαγές ε, στη συνεδρίαση, ε, λόγω και της παρουσίας μεταξύ άλλων και του επιτρέπου Έτιγκερ. Γι' αυτό λοιπόν θα προτιμούσα να περάσουμε ήδη ε, στις ομιλίες των ε, εμπειρογνωμόνων μας. Πολύ ωραία λοιπόν, συμφωνήσαμε ότι ο καθένας θα περιοριστεί σε 10 λεπτά και θα τρέχει και το ρολόι για να το βλέπετε. Και εμένα με βοηθάει αυτό μερικέ φορές. Και το πρώτο, στον πρώτο δίνω το λόγο στον κύριο Οσίτη, ο οποίο είναι από τη ε, Λετωνία. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. <laughs> Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Θα σας παρουσιάσω τις προσδοκίες της περιοχής της Βαλτικής σχέση με την ενέργεια και ορισμένες πτυχές των υποδομών μας και των προτεραιοτήτων τους. Σε ό,τι φορά, όπως αναφέρεται και στα έγγραφα το ε, πρόγραμμα αγοράς ενέργειας της Βαλτικής, BENIP, όπως ονομάζεται. Έχουμε ήδη 40 χρόνια εμπειρίας σε εννέα αλληλοσυνδεόμενα συστήματα ενέργειας με τις δομές της περιφερειακής συνεργασίας και την ε, μορφή συνεργασίας της Βαλτικής που ήδη λειτουργούν. Έκανα κάποια μικρή αλλαγή στις διαφάνειες. κάποιες αλλαγές στο ύφος και στην έμφαση της παρουσίαση. και επίσης κάποιες πρόσθετες πληροφορίες θα δείτε. Εδώ θα δείτε κάτι που βρίσκεται το αντιμετωπίζουν πολλά ευρωπαϊκέ και περιφερειακές αρχές που πρέπει να λάβουν αποφάσεις. Είναι δύσκολο να ληφθούν αποφάσεις, απαιτούν αλλαγές και πρέπει κανείς να σκέφτεται και του μακροπρόθεσμους και του βαχυπρόθεσμου στόχους. Υπάρχουν αρκετά σημεία που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε σχέση με τις υποδομές ενέργειας και τις προτεραιότητές τους. Πολλές από αυτές είναι τεχνικού χαρακτήρα και πρέπει να επιληθούν σε βιομηχανικό και θεσμικό επίπεδο. Ένα σημείο που θέλω να τονίσω και θέλω να σας επισημάνω θα μας απασχολήσει περισσότερο από το δεύτερο και το τρίτο. Δεν θα τα αναπτύξω τόσο γιατί είναι πιο τεχνικά. Στο πρώτο θέλω να σταθούμε. of plan. Για το σχεδιασμό του BEMIP. Βλέπουμε τα πραγματικά αποτελέσματα ως το 2014. Βλέπουμε ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δηλαδή οι διασυνδέσεις των δικτύων της Βαλτικής με τη Σκανδιναβία και τις σκανδιναβικές χώρες. Μιλάμε για εργασίες και έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο είναι σαφές το τι θα συμβεί μετά με τις διασυνδέσεις. That could lead towards... Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε μη εκπλήρωση των δραστηριοτήτων και των δράσεων που προβλέπει το BEMIP. Η δυσκολία εν μέρη οφείλεται στις ιστορικέ ε, ιστορικές σχέσεις εξάρτησης που υπάρχουν με τρίτες χώρες και την υποβάθμιση των υποδομών. Βλέπετε για τις βαλτικές χώρες ότι υπάρχει στενή αλληλεξάρτηση με τα δίκτυα της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Οι χώρες αυτές προφανώς δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε του ΕΟΧ. Επιπλέον άχθος δημιουργεί η περιοχή του Καλίνιγκραντ, που είναι ένας θύλακας της Ρωσίας μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνίας. Τα, τα σύνορά μας με τις ευρωπαϊκές χώρες είναι μόνο το κομμάτι μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας, που είναι πολύ μικρό. Δεν υπάρχουν ακόμη στενοί δεσμοί διασύνδεσης. Επίσης, είναι μια από τις πιο δύσκολες περιοχές απόψη υποδομών της Πολωνίας αυτή. Υπάρχει μόνο ένα καλώδιο υψηλή τάση DC, που συνδέει επίσης την Πολωνία με την Φινλανδία αυτή τη στιγμή. Τα σημεία προσυζήτηση είναι ότι δεν έχουμε πολύ ιστορικό υλικό, τεχνικό υλικό από ιστορικής άποψης. Η επιρροή των τρίτων χωρών θα συνεχίσει να επηρεάζει την εξέλιξη της αγοράς της Βαλτικής για την ενέργεια και την ε, συνεργασία της με την υπόλοιπη Ευρώπη. Για την ασφάλεια της προμήθειας ενέργειας στην όλη περιοχή πρέπει να γίνουν πολλές κινήσεις, διότι αν δεν γίνει τίποτε θα πρέπει να ακολουθήσουμε άλλη πορεία. Goal. Βασικός στόχος λοιπόν είναι να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες απειλές. Η πρώτη απειλή συνεχίζει να υφίσταται. Κατά πρώτον, Έχουμε ένα μονόδρομο της ενέργειας στην αγορά αυτή από την Ρωσία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχέση αυτή θα πρέπει να είναι αμφίδρομη. Έπειτα, δεύτερο σημείο προσεζήτηση είναι οι διασυνδέσεις με το υπόλοιπο των ευρωπαϊκών συστημάτων. Αυτές μπορεί να μην είναι επαρκείς εάν δεν αναπτυχθούν δυνατότητες παραγωγής ενέργειας στις ίδιες τις βαλτικές ε, χώρες. Αυτό οφείλεται στις ανεπαρκείς επενδύσεις στην καλωδίωση που προκαλούνται από διάφορα πρότυπα για το διοξίδιο του άνθρακα, το περιβάλλον και ε, εργασιακά που προκύπτουν από τις τρίτες χώρες, από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Κατά τρίτο, η ενσωμάτωση της βαλτική στην ευρωπαϊκή αγορά μπορεί να μην είναι επιτυχής, να μην είναι πλήρης, διότι επηρεάζεται ιδιαίτερω από τις αγορές εκτός ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου και τη συμπεριφορά των συστημάτων τους. Υπάρχουν πολυάριθμοι πυρηνική σταθμή στην Ρωσία και πολλοί που πρόκειται να χτιστούν στη Λευκορωσία. Προφανώ έχουν διαφορετική συμπεριφορά οι χώρε αυτέ και επηρεάζονται ιδιαίτερω. Επηρεάζουν μάλλον τη δική μας την εξέλιξη, στην ενσωμάτωση αυτή προς την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και την ενεργειακή μας ασφάλεια. Τι προτείνουμε τώρα ζητάτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει ευέλικτες νομοθεσίες και πολιτικές σε ό,τι αφορά τις απομακρυσμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρίτες χώρες. Η ευελιξία, κατά τη δική μου αντίληψη, σημαίνει ότι θα εξεύρουμε κάποιες συγκεκριμένε λύσεις στις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να καλύπτονται και να γίνονται σεβαστές οι ανάγκες ε, συγκεκριμένων απομακρυσμένων χωρών, παραμεθόριων χωρών και περιοχών αυτών των χωρών, ιδίως τις σχέση τους με τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας εάν τυχόν υπάρχουν ερωτήματα. Σας ευχαριστώ που τηρήσατε και το χρονοδιάγραμμα. Πολύ χρήσιμο. Στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Ρομπέρτο Καμπάγιο Γιώχα, ο οποίος είναι επικεφαλής ε, της Ελέκτρικα, της Red Electric από την Ισπανία. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ. να σας συγχαρούμε για το έγγραφο που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο για τη συζήτησή του και για το γεγονός ότι αναγνωρίζετε τις ανάγκες των ενεργειακών δικτύων τα οποία είναι ολοκληρωμένα και αξιόπιστα. Στα θέματα των υποδομών έχουμε προγράμματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος τα οποία θέλουν να μας βοηθήσουν και να εφαρμόσουμε υποδομές προτεραιότητες. Ωστόσο, θεωρούμε ότι αυτή η ανάγκη να υπάρχουν προγράμματα που θα λαμβάνουν υπόψη και το γεγονός ότι είναι ευρωπαϊκή ωφελία. Ε, δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος της διασύνδεσης, διότι εντός των εθνικών δικτύων υπάρχουν και άλλες υποδομές οι οποίες σε μεγάλο βαθμό συνεισφέρουν στη μεγαλύτερη δυνατότητα, δυνατότητα διασύνδεσης ε, στο δίκτυο. Επομένως, τα δίκτυα τα οποία δεν είναι διαμεθοριακά αλλά είναι εθνικά δίκτυα θα πρέπει να ληφθούν ε, δεόντως υπόψη. θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης των ε, ε, υποδομών του TEN-E. Ε, το TEN-E δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί ως συμπίληση των όσων κάνει το κάθε κράτος μέλος, αλλά με ένα όρασμα, όραμα πιο υπερεθνικό, πιο ευρωπαϊκό. Θεωρώ ότι η εμπειρία μας της πρώτης χρονιάς θα πρέπει να βελτιωθεί, ξεκινώντας από τη δεύτερη ε, πρωτοβουλία που υιοθετήσαμε, τα DSO, στους διαχειριστές συστήματος μεταφοράς, για να προχωρήσει αυτό το ε, σχέδιο ανάπτυξης, ε, του δεκαετούς, το δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου πιο αποτελεσματικά. Και νομίζω ότι αυτό περιλαμβάνεται πολύ καλά στο έγγραφο δίνεται μεγάλη σημασία και στις περιφερειακές ε, πτυχές, διότι από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε τη βαθμιδόν ε, δημιουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην ε, νοτιοανατολική περιοχή έχουμε ένα επίπεδο διασύνδεσης με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Εκεί στις περισσότερες περιοχές υπάρχει ενιαία τιμή, τιμολόγηση και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, διότι η Ισπανία και η Πορτογαλία θεωρείται ως ενιαία αγορά σε θέματα διασύνδεσης ενεργειακών δικτύων και αυτό είναι το είδος των πρωτοβουλειών που θα πρέπει να ενισχύσουμε και να, να θεωρήσουμε. Για να είναι δυνατή η πολιτική που θέλουμε, δηλαδή να μην έχουμε πλέον εξάρτηση από τον άνθρακα και να έχουμε περισσότερη εξάρτηση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες για να χρησιμοποιήσουμε ενέργειες οι οποίες ε, είναι δύσκολο να προβλέψουμε σε ασφαλείς ε, συνθήκες, κυρίως ε, σε περιφερειακές χώρες που δεν έχουν τόσο καλές δυνατότητες διασύνδεσης. Και αυτά είναι στοιχεία τα οποία βασίζονται στη διαχείριση της, δι... της ζήτησης ή αποθήκες και δεν ξέρω κάποια στιγμή μπορεί να έχουμε και ηλεκτρικά αυτοκίνητα και να χρησιμοποιούμε όλοι. Ε, αυτές βέβαια είναι πιο μακροπρόθεσμες προοπτικές, αλλά σήμερα το θέμα της ζήτησης, καθώς επίσης και το θέμα των ε, αποθηκών και των ε, χώρων ε, στους οποίους θα μπορεί κάποιος να ε, βρει αποθήκευση ενέργειας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις τεχνικές πτυχές αλλά και τις πτυχές της διαχείρισης και θα πρέπει να ε, σχετίσουμε τις υποδομές για τις μελλοντικέ τους λειτουργίες που γεννιούνται αυτή τη στιγμή. Τη δυνατότητα δηλαδή να λειτουργούν με συνθήκες ασφαλείας και να χρησιμοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. ένα από τα θέματα που τίθεται είναι και το θέμα της κοινωνικής διάστασης και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν και μηχανισμοί οι οποίοι θα πρέπει να εγγυώνται και την δημόσια συμμετοχή, θα πρέπει να συνοδεύονται και από ε, μέσα επικοινωνίας που θα εξηγούν στους πολίτες τη σχέση κόστους-οφελίας αυτών των υποδομών και επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια κάποια εναρμόνιση για τις ε, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Μας ενδιαφέρει σε αυτή τη διαφάνεια να σταθούμε λίγο διότι βλέπουμε και κάποιους διαδρόμους ε, οι οποίοι είναι διάδρομοι προτεραιότητες, ε, κυρίως το διάδρομο ο οποίος φέρνει αιωλική ενέργεια από την Βόρεια Θάλασσα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στην κατασκευή μεγάλων ε, ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Tech, του MedGrid και όλα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν προπομπό του High Grid. Να υπάρχουν δηλαδή δυνατότητες ένωσης των ε, ε, σημείων ε, ανανεώσιμης πηγών ενέργειας από την Αφρική με τις ευρωπαϊκές χώρες. Αφανώς γιατί υπάρχουν πολλές δυνατότητες και επίσης υπάρχουν και φθηνές δυνατότητες ε, αν επενδύσουμε σε τέτοιες σημαντικές υποδομές, αλλά υπάρχει και ένα επιπλέον πολιτικό πλεονέκτημα διότι θα δημιουργηθούν σε περιοχές τις, στις οποίες βρίσκονται οι πηγές ενέργειας και θα δημιουργηθούν υποδομές που σημαίνει ότι θα βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Δεδομένου ότι βιώνουμε και όλα όσα βιώνουμε στη Βόρεια Αφρική είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία και μεγαλύτερη ε, συμμετοχή στα ενεργειακά ζητήματα και αυτό φαίνεται σε προγράμματα όπως αυτό. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα από τα πρώτα βήματα για να αναπτύξουμε αυτές τους μεγάλους ε, διαδρόμους ηλεκτρικής ενέργειας που θα βοηθήσουν τόσο τους πολίτες των χωρών προέλευσης των ενεργειακών πόρων, όσο και τους πολίτες που θα καταναλώσουν αυτή την ενέργεια, η οποία θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε τον ορισμό του διαδρόμου θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λειτουργούν αυτοί και θα πρέπει να υπάρχει και συντονισμός με τα σχέδια ανάπτυξης επιτόπου. Υπάρχουν δυνατότητες ε, διασύνδεσης, ε, οι οποίες στην ε, περίπτωσή μας μας φαίνονται ότι είναι ήπιες. Θα πρέπει να υπάρχει ως ελάχιστο 6.000 ΜΒ με την Γαλλία ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε 4.000 μόνο και αυτά τα γνωρίζετε, γνωρίζετε ότι υπάρχει διασύνδεση από τα Πυρηναία και θα πρέπει να υπάρχει και διασύνδεση υποθαλάσσια στον ε, Βυσκαϊκό κόλπο. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι το θέμα της ε, χρηματοδότησης και των μέσων χρηματοδότησης. Θεωρώ ότι αυτά αναφέρονται παρκώς ε, στη συνθήκη, διότι αυτά τα προγράμματα υποδομών είναι πολύ περίπλοκα από τεχνική σκοπιά και επιπλέον είναι και διαμεθοριακά. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ε, χρηματοδότηση, ίσως και σταδιακή, δεδομένου ότι ορισμένες φορές υπάρχει και μια κάποια βεβαιότητα σε αυτές τις υποδομές και αυτό που είναι πολύ σημαντικό ώστε κατά κάποιο τρόπο να διασφαλίζεται και η ε, η υποστήριξη των ε, TSOs, ε, των διαχειριστών συστημάτων μεταφορός, είναι να υπάρχουν ρυθμιστικά πλαίσια τα οποία θα είναι σταθερά και ελκυστικά και θα μας επιτρέπουν να έχουμε και ανταγωνιστικές τιμές. Θα μπορούσαμε ίσως να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει και νομοθετική πρόταση μέσω μιας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, προσωμείωση του κόστους. Ίσως ε, ε, να γίνει κάτι τέτοιο προβλέπεται για τον Ιούνιο του 2011 και θα πρέπει εμείς να δώσουμε και όθηση προς αυτή την κατεύθυνση. Οι τρεις-τέσσερις μορφές τιμολόγησης που θα μπορούσαμε να έχουμε ε, η, με των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς για να λάβουν υπόψη τους μηχανισμούς αποζημίωσης, τα τιμολόγια ε, και ούτω καθεξής θα πρέπει να αναθεωρηθούν διότι αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός που διαθέτουμε δεν είναι ικανοποιητικός ε, και δεν είναι αυτός που χρειαζόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε μηχανισμούς αποζημίωσης για τις περιοχές οι οποίες πλήττονται λόγω της ανάπτυξης των, ε, της διαθήκης, αλλά επίσης και για υποδομές που επειδή ακριβώς ε, δεν είναι διαμεθοριακή διασύνδεση αλλά εσωτερικό δίκτυο, μας επιτρέπουν να αυξήσουμε τις δυνατότητες διασύνδεσης. Χρειαζόμαστε λοιπόν μέτρα και συγκεκριμένες προθεσμίες για να τηρήσουμε αυτά τα όρια. Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετική ιδέα το One Stop Shop, αυτή η ενιαία ε, θηρίδα. Και είναι πολύ λογικό το ότι θα πρέπει να υπάρχουν και οικονομικά κίνητρα σε περιοχές ε, όπου ε, οι αδειοδοτήσεις απαιτούν παρακολούθηση. Θα πρέπει να θεωρηθούν αυτά προγράμματα προτεραιότητα σε συγκεκριμένα εθνικά δίκτυα, τα οποία μπορεί να έχουν και ε, επιπτώσεις στα νοριακές περιοχές και πρέπει να λάβουμε υπόψη το ενίο σύστημα όπως έχουμε για παράδειγμα στην Πορτογαλία με την Ισπανία και το γεγονός ότι ο στόχος διασύνδεσης με την, Ισπανία, με την Γαλλία θα πρέπει να αυξήσει τη δυνατότητά του τουλάχιστον μέχρι τα 6.000 ΜΒ, ε, αν όχι και τα 10.000 που θα ήταν ο πιο λογικός στόχος. Ένα σημείο που είναι εξίσου σημαντικό είναι να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα μηχανισμό ολοκλήρωσης εάν δεν υπάρχουν και δυνατότητες αποθήκευσης και επίσης θεωρούμε ότι οι TSOs θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες της, ε, των εγκαταστάσεων διασύνδεσης διότι έτσι θα έχουμε μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική αποδοτικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Äh, Επόμενος, κάλευ Στάντιος, ε, είναι από την ε, ABB Smart Grids. Και είναι, νομίζω είναι η δική σας η σειρά. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το δικό μου το θέμα είναι η ανάπτυξη των ε, Smart Grid. των ευθειών δικτύων. Ας δούμε λοιπόν ε, τι ακριβώς έκανε ο Διεθνής Οργανισμός μέχρι το ε, τι θα κάνει μέχρι το 2030 και προβλέπετε ότι η ε, προσφορά θα ξεπεράσει τη ζήτηση. Η υποδομή για της, ε, για την ενέργεια είναι από τους μεγαλύτερους τομείς επενδύσεων και πάνω από το 50% των επενδύσεων είναι στο δίκτυο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι ανανέωση των υφιστάμενων δομών και στον υπόλοιπο κόσμο νέες κατασκευές. Πρόκειται λοιπόν για μια μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία για πάρα πολλέ ευρωπαϊκές εταιρείες. Όσον αφορά το FES δίκτυο, είναι ένα σημαντικό στοιχείο για ένα βιώσιμο ε, σύστημα ενέργειας γιατί αυξάνεται, βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα, βελτιώνεται το ποσοστό των ανώσιμων πηγών ενέργειας και παρόλα αυτά παραμένει ιδιαίτερα αξιόπιτο το FES, το FES δίκτυο. Ε, βασικές προκλήσεις ε, είναι η ενσωμάτωση ανανώσιμων πηγών ενέργειας και η ενέργεια, η ε, κατανομή της ενέργειας στο δίκτυο. Οι ενεργοί καταναλωτές επιθυμούν να αμείβονται για την ε, ισχύ που ε, προσφέρουν και για την immobility. Είναι περισσότερο βασικό φορτίο στην ενέργεια. Επίσης, αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι η κατανάλωση όταν υπάρχει ε, ενέργεια που περισσεύει, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την περισσεύουσα ενέργεια για να αποφευθούν οι ώρες ε, της εχμής. Βέβαια, αυτό απαιτεί κίνητρα για τους καταναλωτές ε, που σημαίνει ότι τα εφή δίκτυα δεν είναι μόνο ένα τεχνικής φύσεως θέμα, αλλά είναι επίσης και ένα θέμα που έχει σχέση με τα επιχειρηματικά μοντέλα και με το ρυθμιστικό πλαίσιο οι περισσότερες προκλήσεις ε, βρίσκονται στο ποσοστό ε, κατανομής σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητο ε, να υπάρχει ένα τέτοιο ευφυές δίκτυο για να υπάρχει και η μέγιστη χρήση της νόσων των πηγών ενέργειας. Έτσι λοιπόν για να έχουμε τεχνικής φύσεως λήξης, για να μελτήσουμε τα συστήματα, να έχουμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, να προσαρμόσουμε τα ρυθμιστικά μοντέλα και να τα στηρίξουμε, το καθήκον μας είναι ε, να εμπλέξουμε όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Οι προκλήσεις που υπάρχουν για συνεργασία ανάμεσα στους οργανισμούς κοινή ωφελία και τους παρόχους ενέργειας, τις μεγάλες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ερευνητές και όσους αναπτύσσουν πολιτική, όλα αυτά απαιτούν να υπάρχουν ένα FES δίκτυο, το οποίο καθίσταται ένα σημαντικό στοιχείο που στηρίζει τη βιομηχανική ανάπτυξη. Δύο παραδείγματα βλέπουμε εδώ, τα οποία αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή. Είναι το ε, λιμάνι της ε, Στοκχόλμης, ε, και ένα ευφυές e δίκτυο στο Γκότλαντ, το οποίο εστιάζεται στην ενσωμάτωση μεγάλων ποσοτήτων ανέμου στο δίκτυο ε, διανομής. Όσον αφορά το FES δίκτυο, πρόκειται για μια παγκόσμια έννοια, όμως ε, αναμφισβήτητα με τοπικούς χάρτες πορείας. Είναι διαφορετικές οι προκλήσεις στα διάφορα μέρη του κόσμου, γιατί έχουμε και διαφορετικές χώρες. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να υπάρχουν και μεμονωμένα προγράμματα. Ε, τα νομικά και τα άλλα εμπόδια πρέπει να αρθούν και πρέπει να προσφέρονται κίνητρα έτσι ώστε ε, οι ε, χορηγοί και οι πάροχοι να ενθαρρύνονται να επενδύουν στο FES δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή αγορά, αυτό, αυτή αναπτύσσεται. Βέβαια οι ε, παραγωγοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν και την τελευταία τεχνολογία. Εξάλλου, το, πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πρέπει και αυτό να συζητηθεί. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρχει ε, μια ενεργός διαδικασία παρακολούθησης όλων των τοπικών πρωτοβουλειών. Το FTS δίκτυο, όπως αναφέρθηκε, για να μπορέσουμε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν, να έχουμε μια νέα ε, αγορά, πρέπει να ορίσουμε και τους μηχανισμούς πώς μπορεί να λάβει η χώρα η καινοτομία. Η δημιουργία και η υποστήριξη, η οικονομική υποστήριξη αυτών των ε, καινοτομιών, έρευνας και τεχνολογίας είναι ένα πολύ σημαντικό καθήκον που πρέπει να χρηματοδοτείται. Τώρα, το πώς αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να ε, συνδεθούν με την έρευνα, αυτό ε, μπορεί να γίνει μέσα από την ιατρική e Energy, ένα δίκτυο που δημιουργείται αυτή τη στιγμή. Οι δυνατότητες που προσφέρει το FES δίκτυο οι δυνατότητες αυτές είναι πολύ σημαντικές για τις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Στην Ευρώπη ε, είμαστε σε καλή θέση, μπορούμε να λάβουμε ηγετικό ρόλο και να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον τομέα που προσφέρετε. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ε, σας ευχαριστούμε θερμά και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον δόκτωρα Εκατρόστα, ο οποίος είναι μηχανικός και έχετε το λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή που κάνατε. Θα ήθελα επίση να προσθέσω ότι εμεί ασχολούμεθα κυρίω ε, με την ενσωμάτωση στο δίκτυο των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Όχι μόνο με γεννήτριες αιωλική ενέργειας. Ε, και θα ήθελα ε, να σας παρουσιάσω την Ευρωπαϊκή Μελέτη Δικτύων. Έχετε ερώτημα? Α, όχι, διακόπτη μελητής. Όχι, όχι, όχι, συνεχίστε. Κοιτάξτε, <laughs> τα μέλη ζητάνε το λόγο πριν μπουν στην αίθουσα. Αν συνηθίστε σε αυτό, γίνεται στο Κοινοβούλιο. Έχουμε λοιπόν μία μελέτη που θα σας την παρουσιάσω είναι μια μελέτη ε, που αφορά το χρονικό διάστημα και μέχρι το 1950. Και αυτό που ενδιαφέρει είναι το εξή. Ε, η ε, Greenpeace παρουσίασε ένα σενάριο, πανεστατικό σενάριο για την ενέργεια που ίσως να το γνωρίζετε. Και γενικά λοιπόν δεν λαμβάνονται υπόψη δυστυχώς οι υποδομές δικτύων. Αυτό λοιπόν ήταν το δικό μας το καθήκον να κάνουμε τη σχετική μελέτη και γι' αυτό καταρτήσαμε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο δικτύων. Επίσης, να πω το η προσέγγιση μας ε, ήταν αφενός ε, να ελέγξουμε τον εφοδιασμό, ασφάλεια εφοδιασμού. Ε, ελέγξαμε τελευταία 40 χρόνια τις κλιματικές συνθήκες, επιλέξαμε ακραία καιρικά φαινόμενα και κατόπιν εξετάσαμε επίσης τι μπορεί να γίνει με την ενσωμάτωση των ανώσιμων πηγών ενέργειας. Και αυτά τα κάναμε για ένα ολόκληρο χρόνο. θεωρήσαμε, η στόχος ήταν μέχρι το 2030 περίπου το 70% ε, της ενέργειας να είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι τότε να έχουμε φύγει από την πυρηνική ενέργεια, να μην υπάρχει κανένα πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη ε, και να μην χρησιμοποιείται και σχεδόν καθόλου ο άνθρακας. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα κατά πόσον αυτό είναι δυνατό να γίνει. Ε, Τέτοιο αυτό ερώτημα και εμείς κάναμε τη σχετική έρευνα. Βεβαίως ένα θέμα που ενδιαφέρει είναι το εξής. Αν εξετάσει κανείς μόνο τις ε, προτεραιότητες ε, ε, και προτεραιότητα δώσει στις ανώσιμες πηγές ενέργειας και πει ότι αυτές προηγούνται στο δίκτυο και διασυνοριακά, μπορεί κανείς να πετύχει πάρα πολλά χωρίς να χρειαστεί ε, να ε, κάνει μεγάλες αλλαγές στο δίκτυο. Ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω είναι το εξή ερώτημα. τι ακριβώς μπορώ να πετύχω με την επέκταση των δικτύων και επίσης και με την αποθήκευση ενέργειας. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι με την επέκταση δικτύων μπορούμε να επιτύχουμε πάρα πολλά και μάλιστα με προσιτό κόστος. Άρα δηλαδή εδώ μπορούμε να επηρεάσουμε την ε, ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και να ασκήσουμε θετική επιρροή στον, ε, στην ασφάλεια εφοδιασμού. Μπορεί να αυξηθεί λοιπόν η ασφάλεια εφοδιασμού και διαπιστώνουμε ότι οι καταστάσεις ε, ε, όπου για αρκετές ημέρες δεν έχουμε αιωλική ενέργεια, παρήματο χάρη ε, στη Βόρεια Θάλασσα, εκεί με αποθηκευμένη ενέργεια μπορούμε να ε, συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Η επέκταση των δικτύων, όπως ακούσαμε, είναι κάτι που προποθέτει ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό και γι' αυτό έχει και κάποιους περιορισμούς. Το δίκτυο το οποίο ε, σχεδιάσαμε για το 2030 δείχνει ότι πρέπει να υπάρξουν πολλές αναβαθμίσεις και ως εκ τούτου πράγματι ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να το βελτιστοποιήσουμε και να επεκτείνουμε τις υπάρχουσες δομές. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τη νότια προς την κεντρική Ευρώπη. Εκεί είναι απαραίτητο να υπάρξουν ε, ουσιαστικές ε, ουσιαστικές διασυνδέσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη Βαλτική θάλασσα. Ε, μέχρι το 2030 θα χρειαζόμαστε 100.000 χιλιόμετρα και η επένδυση θα είναι περίπου 70 δις ευρώ. Ε, αυτό λοιπόν θα μπορούσε να είναι ένα super grid ε, μέχρι το 2030 το οποίο θα αφορά κυρίως τον άξονα βορρά-νότου ε, και το ε, εξωχώριο δίκτυο. Και το 2015 θα είναι αυτή η κατάσταση που βλέπετε στη διαφάνεια. Μέχρι το 30 δεν θα έχουν γίνει πολλές επενδύσεις. αλλά μέχρι το 2050 θα μπορούμε να να έχουμε στην Ευρώπη μέχρι και 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, βεβαίως ε, οι επενδύσεις είναι πολύ σημαντικές, ε, υψηλής κλίμακας και πρέπει να γίνουν και απαραίτητες προσπάθειες στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας. Ανακεφαλώνοντας λοιπόν θα ήθελα να πω το εξής. Η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να είναι από τις πρώτες προτεραιότητες σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλουμε να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες ε, στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας ε, ενέργεια που δεν καταναλώνεται δεν πρέπει και να παράγεται αλλά ούτε και να μεταφέρεται. Επίσης ε, πρέπει να κατασκευαστούν καινούργιοι αγωγοί και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρχει ε, βελτιστοποίηση αυτών των αγωγών και να υπάρξει και χρήση των υφιστάμενων δομών. Όσον αφορά τη διαχείριση και την αποθήκευση, εκεί τα ευφύ δίκτυα θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί υπάρχουν περιορισμοί στην επέκταση των υφιστάμενων δικτύων. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με την απαιτούμενη ταχύτητα με βάση τι ανάγκε μα. Και τέλο, το FES δίκτυο, Electricity Highways, ε, το ακούσαμε αυτό. Αυτά είναι απαραίτητα για να έχουμε έχουμε μια Ε, ίση κατανομή της ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και εάν γίνουν όλα αυτά, τότε μέχρι το 2030 θα μπορούμε να μεταπηδήσουμε σε ένα άλλο ε, δίκτυο το οποίο θα βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο αέριο. Αέριο γιατί εκεί χρειαζόμαστε ε, ευέλικτες ε, εγκαταστάσεις όπου θα υπάρχει και συνδυασμός με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το αέριο εάν τελικά υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας ε, στον τομέα της ε, θερμότητας, ε, τότε η κατανάλωση αερίου δεν θα αυξηθεί σημαντικά. Κατά τη δική μας λοιπόν άποψη είναι σημαντικό να γίνουν και άλλες έρευνες και κατόπιν τούτου ε, θα πρέπει τα ε, ευρωπαϊκά στοιχεία περιδικτύων να είναι δημόσια προϊστά σε όλους για να μπορούν να γίνουν και οι απαραίτητες μελέτες. Εάν έχετε ερωτήσει, παρακαλώ, ευχαρίστω είμαι στη διαθεσία να απαντήσω. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος, και ευχαριστούμε και όλους τους ε, συναντέλφους σας και χαίρομαι πάρα πολύ για το πόσο πιστά τηρείτε το χρόνο σας. Και αυτό ε, θα μας βοηθήσει για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Είναι μεγάλη μου τιμή να μπορώ να μιλήσω σήμερα στην Επιτροπή σας. Είμαι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπεύθυνου Φορέα για την Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της δημοκρατία της Τσεχίας. Η, δημοκρα... η βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας έχει μεγάλη ιστορία στην Δημοκρατία της Τσεχίας και είναι ένα ενοποιημένο σύστημα που σκοπό έχει να καλύπτει τις ανάγκες όλων των πελατών. 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες την εβδομάδα, την, το έτος, συγγνώμη, με λογικές τιμές. Θα δείτε ότι υπάρχουν έγγραφα που περιγράφουν την κατάσταση της τελευταίας δεκαετίας και έχουν δημοσιευτεί και το θέμα είναι κατά πόσον πραγματικά καταφέρνουμε το στόχο της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ε, στο βαθμό που όλοι τον χρειάζονται. Αυτό δεν περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Για το 2009 και μόνον η ασφάλεια της παροχής ε, συζητήθηκε σε βαθμό μικρότερο από αυτόν που χρειαζόταν. Επίσης, οι στόχοι για την ηλεκτρική ενέργεια άνθρακα που παράγεται από ανανόσιμε πηγέ ενέργεια δεν ε, αναλύονται αρκετά στα συγκεκριμένα έγγραφα. Εδώ λοιπόν ωστό, το ερώτημα είναι μήπως έχουμε καταλήψει το βασικό μας στόχο να παράσχουμε ηλεκτρική ενέργεια σε όλους ανεξαιρέτως. Όχι είναι η απάντηση. Δεν έχουμε καταλήψει το στόχο αυτό. Πρέπει να έχουμε υπόψη το γεγονός ότι ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας πάντοτε λειτουργούσε ενιαία. Είναι δύσκολο να αποθηκευτεί ενέργεια και είναι δύσκολο να βρίσκεται πάντα τη σωστή ισορροπία μεταξύ ζήτηση και προσφορά. Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση καθορίζει πόση ενέργεια παράγεται. Δηλαδή, βασιζόμαστε σε μια απλή αρχή τη φυσική ε, για την βιομηχανία τη ηλεκτρική ενέργεια στην Τσεχία. Όταν όμω μιλάμε για νεώσουμε πηγές ενέργεια δεν καθορίζει η ζήτηση την παραγωγή, αλλά η διαθεσιμότητα των πόρων. Δηλαδή, κατά πόσον υπάρχει ηλιοφάνεια και άνεμος. Ας σκεφτούμε όμως πιο απλά τα πράγματα. Όλη στη ζωή σας θα έχετε χρησιμοποιήσει ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Έχετε αναρωτηθεί όμως τι είδους ηλεκτρικά εργοστάσια προτιμάτε. Πιστεύετε ότι γύρω σας αυτό το ερώτημα έχει τεθεί αρκετά. Να σας δώσω λίγα, ε, κάποια παραδείγματα. Η ηλιακή ενέργεια λόγου χάρη και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια. Μπορούμε να πούμε ότι είναι φιλική προς το περιβάλλον, μπορούμε να, να πούμε ότι καλύπτει αυτή τη βασική μας αρχή. Ή τα εργοστάσια υδροελεκτρικής ενέργειας. Και αυτό φαίνεται μια καλή ε, λύση, όμως τα φράγματα δεν αρέσουν πολύ σε όρους. Τα εργοστάσια πυρηνική ενέργειας μετά από όσα έγιναν στην Ιαπωνία βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να τα προκρίνουμε ως επιλογή. Ε, άλλου είδους ε, παραγωγή ενέργειας ίσως. Η ηλιακή λοιπόν ενέργεια και οι ηλιακές καταστάσεις ποτέ δεν θα καταφέρουν να μας δώσουν τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που χρειαζόμαστε. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες τεχνικού χαρακτήρα, διότι θα σας δυσκόλευα, θα μπορούσα να μιλήσω για τα σύντομα κυκλώματα, για διάφορους τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά θα περιοριστώ στα εξή. Στον τομέα μας έχουμε εμπειρογνώμονες που τους άλλως θα καλύψουν τις τεχνικές λεπτομέρειες. Για μας η βασική πρόκληση είναι να καλύψουμε την ποιότητα της παροχής. Ας δούμε τι γίνεται με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Φαντάζομαι όταν ρωτάτε τους ανθρώπους για τα καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας ε, θα σας απαντήσουν δεν μας αρέσουν. Χαλάνε το τοπίο, είναι άσχημα, ε, δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ε, προκαλούν κινδύνους και απειλούν την υγεία. Πολλέ φορέ λένε εντάξει, αλλά δεν τα θέλω στο δικό μου το σπίτι, στη δική μου τη γειτονιά. Συζήτησα με συναδέλφου από άλλε ανάλογε εταιρείε και μα είπαν ότι παρόμοιε απαντήσει λαμβάνουν. Σε όλη την Ευρώπη τα ίδια προβλήματα προκύπτουν. Όμω ο καθένα θέλει πρόσβαση στον ηλεκτρισμό διαρκώ, συνεχώ. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε το θέμα σε δημόσια διαβούλευση. Δηλαδή, πώς θα παρέχουμε ηλεκτρική ενέργεια σε όλους. Βασικό στρατηγικός στόχος για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι ακριβώς αυτός και για τα κράτη-μέλη. Να διασφαλίσουμε επαρκέ ποσό ηλεκτρισμού για όποιον το χρειάζεται επαρκέ ποσότητε ηλεκτρική ενέργεια. Καλή ποιότητα ηλεκτρική ενέργεια 24 ώρε το 24ωρο και 365 μέρε το χρόνο όπω είπα προηγουμένω. Ήθελα λοιπόν εδώ να προτείνω ένα νέο στρατηγικό στόχο για να προετοιμάσουμε το σύστημα ηλεκτρική ενέργεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψει τον φιλόδοξο στόχο του ποσοστού χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια που έχουν ε, τεθεί για το ενεργειακό μα μείγμα τα συστήματα μεταφοράς δεν είναι ακόμη απολύτως έτοιμα για τις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Εάν ετοιμαστούν θα πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτή τη στιγμή τα συστήματα μεταφοράς και μετατροπής χρειάζονται ακόμα πολλέ εργασίες για να αξιοποιήσουν τη νέα ενέργεια από τις ανανεώσιμε πηγές. Δεν μπορούμε να τα πετάξουμε όμως τα συστήματα αυτά, πρέπει, πρέπει κυρίως να τα ανανεώσουμε. Και αυτό γιατί δεν αρκεί να πλουστεύσουμε μόνο τις διαδικασίες, πρέπει και να επιταχύνουμε το σύστημα εξουσιοδοτήσεων και αδειοδότησης. Συνήθως χρειάζεται τουλάχιστον μια δεκαετία για να λάβει κανείς εξουσιοδότηση. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Αν δεν γίνουν αλλαγέ, θα υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Επόμενος, ε, η επόμενη, η κυρία Τσερλίκοβα η οποία είναι στέλεχος, ε, ασχολείται με επενδύσεις ε, στον τομέα του αερίου. Σιγά σιγά λοιπόν ε, περνάμε τώρα πλέον στο αερίο και θα ακούσουμε δύο εμπειρογνώμονες για το θέμα. Το κυρία Τσιρλίκοβα, παρακαλώ έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ, διότι δίνετε τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς ε, Φυσικού Αερίου να σας απευθύνει το λόγο για την ανάπτυξη των υποδομών, διότι εσείς ε, υποστηρίξατε τη δημιουργία αυτού του οργανισμού μέχρι, μέσω του τρίτου πακέτου νομοθεσίας για την ενέργεια. Και επομένως ο οργανισμός μας συμμετέχει ιδιαίτερα στην ανάλυση των επενδύσεων που χρειάζονται υποδομές σε βράχη και μακροπρόθεσμα. Η Έντσογκ αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί 33 διαχειριστές συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου από 23 χώρες. Πριν περάσω στη συνεισφορά του, της ΕΝΤΣΟΚ για την ε, δημιουργία υποδομής για ε, τις προτεραιότητες. Ε, θα σας πω κάποια πράγματα για τα θέματα τα οποία επισημάνονται στην πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προτεραιότητες της υποδομές. Εάν αναφερθούμε στην ανάπτυξη της υποδομής για το μέλλον, η προτεραιότητα είναι κυρίως να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο, ολοκληρωμένο και ισχυρό δίκτυο είναι εξαιρετικά σημαντικό να βρούμε κοινό επίπεδο συνεννόησης για το τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο κατάλληλο. Κατάλληλο σημαίνει για μας κάτι το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την αγορά. Ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την ασφάλεια εφοδιασμού, ε, συμπεριλαμβανομένε και τις διαφοροποιήσεις του εφοδιασμού, που σε κάποιες ε, περιπτώσεις μπορεί να συνεπάγεται και πολιτικές λύσεις, αλλά οι πολιτικές λύσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τις ε, ρεαλιστικές δυνατότητες προμήθειας και την αντιγωνιστικότητα του φυσικού αερίου. Επιπλέον, εάν αναφερθούμε στην υποστήριξη της ανάπτυξης αυτής εντοπίζοντας προγράμματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποφύγουμε την ε, διάκριση μεταξύ ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Τέλος, κατ' εξίσου σημαντικού, ε, κατάλληλο θα πρέπει επίσης να σημαίνει και βιώσιμο για τους εθνισμένους διαχειριστές ε, συστημάτων όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και τη ρύθμιση, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάντα. Και εδώ ερχόμαστε στο ρόλο του εθνικού ρυθμιστή. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε το κατάλληλο ολοκληρωμένο αξιόπιστο ευρωπαϊκό δίκτυο χωρίς να υπάρχει και εθνική νομοθεσία η οποία θα εναγκαλίζει το ευρωπαϊκό όραμα. Και αυτό φυσικά αφορά κυρίως ε, τις τιμολογήσεις που χρησιμοποιούνται στην εθνική νομοθεσία για την ε, ρύθμιση των ε, μονοπωλίων. Αυτά τα οποία καθορίζονται στο τρίτο πακέτο ενέργειας για τους μηχανισμούς ε, κινήτρων θα πρέπει να εφαρμοστούν το δίχως άλλο. Την περασμένη εβδομάδα σε μία διάσκεψη υπήρχαν τρεις εκπρόσωποι από τρεις διαφορετικές εθνικές ρυθμιστικές αρχές οι οποίοι δεν κατάφεραν να μα πούν τι μηχανισμούς ε, κινήτρων θα εισαγάγουν προκειμένου να εφαρμόσουν το τρίτο πακέτο ε, ενέργειας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό. Όσον αφορά τώρα τη μακροπρόθεσμη ε, ρύθμιση των υποδομών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το νέο περιβάλλον το οποίο θα δημιουργηθεί μέσω των δικτύων και των κατευθυντηρίων γραμμών πλαίσιο, διότι οι νέοι κανόνες θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις ε, για το ποια υποδομή χρειαζόμαστε. Επομένως, η εθνική νομοθεσία είναι ουσιαστική για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου δικτύου φυσικού αερίου, που το οποίο θα υποστηρίξει το μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό όραμα για την ε, αγορά ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει και μία σειρά από διευκολύνσεις ε, για την ανάπτυξη του δικτύου. Να σας πω λίγα πράγματα για την άποψη των ε, TSOs για το φυσικό αέριο, για, αυτό το νέο, για αυτούς τους νέους μηχανισμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την περιφερειακή συνεργασία και κατανοούμε απολύτως γιατί ενδιαφέρεται. Από προσωπική πείρα θα ήθελα να σας επισημάνω ότι η υποχρεωτική περιφερειακή συνεργασία μπορεί να μην μας δώσει πάντα τα αναμενόμενα αποτελέσματα εάν δεν έχουμε ένα σαφές όραμα του στόχου μας και των κοινών ωφελών για τους λόγους για τους οποίους όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εμπλακούν στη διαδικασία. Διότι ο καθένας μπορεί να αντιλαμβάνεται διαφορετικά ε, τις, ε, ε, τα ωφέλη σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν ο ρόλος και οι υπευθυνότητε για όλους τους ενδιαφερομένους θα πρέπει να καθοριστούν σαφώς και θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων. Όσον αφορά τον εξορθολογισμό των ε, διαδικασιών αδειοδότησης, είναι πολύ σημαντικό οποιαδήποτε νέα νομοθετική πρόταση να μην δημιουργεί ε, προγράμματα δεύτερης κατηγορίας διότι κάποιο μικρό πρόγραμμα εθνική στρατηγικής σημασία μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για να ε, υπερτονίσει τα ωφέλη ενός προγράμματος που μπορεί να είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Και στην περίπτωση που στην οποία υπάρχει διαφορετική μεταχείριση για το μικρότερης κλίμακας ε, πρόγραμμα μπορεί να καθυστερήσει και συνεπώς τα ωφέλη μπορεί να μην υπάρχουν. Και ε, θα λείπει κάτι από το πρόγραμμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Αυτό φυσικά ισχύει και για τα μικρότερα ανταγωνιστικά προγράμματα, διότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν και εναλλακτικέ λύσεις ε, για τα μεγαλύτερα προγράμματα υποδομών που στις περισσότερες περιπτώσεις ε, προσελκύουν όλη την προσοχή μας. Ένα άλλο εργαλείο το οποίο αναφέρεται το οποίο θεωρείται ένας καλός τρόπος για να προοδεύσουμε, είναι ε, το εργαλείο της κατανομής του κόστους. Ίσως θα μπορούσε να μας βοηθήσει να επιλύσουμε κάποια θέματα και νομίζω ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου σε αυτή την περίπτωση. Αυτό όμως που έχει περισσότερη σημασία είναι να εφαρμόσουμε το μηχανισμό κινήτρων που σας ανέφερα και προηγουμένως, διότι εμείς θεωρούμε ότι εάν εφαρμοστούν καταλήλως οι μηχανισμοί κινήτρων, η ανάγκη ενός ειδικού εργαλείου κατανομής κόστους ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη, τουλάχιστον για τον τομέα του φυσικού αερίου. Όσον αφορά τα νέα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, εμείς χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία αλλά θεωρούμε ότι μια ανάλυση των μακροπρόθεσμων συνεπειών στην ανάπτυξη της υποδομής θα πρέπει να αξιολογηθεί πολύ προσεκτικά. Θα πρέπει να δούμε τι θα αλλάξει εάν έχουμε ρυθμισμένους και μη ρυθμισμένους φορείς και τα έργα, κυρίως για τους ε, ρυθμισμένους ε, διαχειριστές συστημάτων μεταφορών, δεν θα πρέπει να τιμωρούνται όταν θα χρησιμοποιούν τέτοια νέα καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης. Ίσως δεν θα πρέπει να βιαστούμε και να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε ποια θα είναι αυτά τα μέσα, διότι αν ε, υπάρχουν οι μηχανισμοί κινήτρων, μπορεί οι ανάγκες ε, για να έχουμε νέα καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης να μην είναι ίδιες. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, αλλά θα ήθελα να σας ε, δείξω τι ακριβώς κάνει ο ένσοκ. Για να σηματοδοτεί την αγορά τι ακριβώς ε, χρειάζεται από πλευράς υποδομής. Έχουμε το δεκαετές ε, πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου και έχει δημοσιευθεί. Είναι το πρόγραμμα το οποίο αφορά την επόμενη δεκαετία ε, και από την Πέμπτη θα ξεκινήσει και μια διαδικασία διαβούλευσης ε, επί του προγράμματος. Πρόκειται για μια πολύ εύρωστη ανάλυση των υποδομών φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αξιολογεί και την ε, τις δυνατότητες του ε, δικτύου για ε, ε πολυάριθμα ε, σε εναλλακτικές εκδοχές. Αν χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας ή μπορείτε να συμμετάσχετε και στο workshop που θα γίνει την Πέμπτη. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταίος στο πρώτο πάνελ ο κύριος Ζαν Τσάνταμ, ο οποίος είναι πρόεδρος ε, του Διοικητικού Συμβουλίου της Πολωνικής LNG. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση και τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω την άποψη της βιομηχανίας. Εγώ εκπροσωπώ την Gas System, την ε, πολωνική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας που είναι τελείως ε, αποσυνδεδεμένη και τελείως ανεξάρτητη. Στην παρουσίασή μου σε αυτό το πολύ προχωρημένο έγγραφο θα μιλήσω πολωνικά. Οπότε από, από τώρα βάλτε τα ακουστικά σας. Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας πω ποια είναι η δική μας άποψη για την ηλεκτρική ενέργεια στην κεντρική Ευρώπη. Εάν δείτε αυτό, αυτή τη διαφάνεια θα καταλάβετε ότι όλες μας οι πηγές προμήθειας πηγαίνουν από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Εδώ δηλαδή υπάρχει ένα φαινόμενο μονομέρειας. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια σαφή στάση από την άποψη της παροχής και μια σαφή στάση από την άποψη της εξάρτησης. είδαμε σε καταστάσεις κρίσης να υπάρχει πάυση παροχής του φυσικού αερίου. Συνέβη το 2006 ήδη. Και στην αγορά μας βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ οι περιορισμοί, είναι περιορισμένη η αγορά μας και ξέρετε ότι η αγορά αυτή αφορά την Πολωνία, την Αυστρία, την ε, Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία με συγκεκριμένους καταναλωτικούς κινδύνους. Άλλη είδους επέσεις κατανάλωση σε σχέση με αυτό που καταναλώνουν λόγω χάρη άλλες ομάδες χωρών όπως τις Μπενελούξ. Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις χώρες χρησιμοποιείται ως πηγή παραγωγής ενέργειας σε μεγάλο βαθμό ο άνθρακας. Και αυτό έχει ριζώσει βαθιά στην οικονομική διαχείριση των συγκεκριμένων χωρών. Ο τρόπος που λειτουργούμε έχει καθοριστεί από αυτή τη συμπεριφορά. Δημιουργούνται λοιπόν συνθήκες που δεν επιτρέπουν την άμεση εκδίπλωση μιας ε, όριμης αγοράς φυσικού αερίου. Αν και κάτι τέτοιο ξέρουμε ότι επιδιώκεται, θα βοηθούσε πολύ την ανάπτυξη του δυναμικού της κεντρικής Ευρώπης. Όμως υπάρχουν στοιχεία που αφορούν την ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επηρεάζουν τη δική μας αγορά. Λόγω χάρη η πολιτική για τις κλιματικές αλλαγές της, Ευρω... της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι στόχοι για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και το δυναμικό παραγωγής φυσικού αερίου όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής. Εδώ πρέπει να δούμε πόσο μπορούμε να έχουμε εργοστάσια που θα λειτουργούν με φυσικό αέριο και γενικότερα ποια πολιτική παροχής ενέργειας ακολουθούμε. Πώς στηρίζονται κάποια προγράμματα που θα μπορούσαν να εξαλείψουν τις ενεργειακές νησίδες και προγράμματα όπως το ΜΙΠ ή ο διάδρομος Βορρά-Νότου. Αυτή είναι η απάντηση του εθνικού μας φορέα στις διάφορες προκλήσεις που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στις ενεργειακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ασχοληθεί ιδιαιτέρως τα τελευταία δύο χρόνια στο να δημιουργήσουμε τις κατάλληλε υποδομέ για το φυσικό αέριο στην Πολωνία και γενικότερα στην κεντρική Ευρώπη. Έχουμε δύο μεγάλα προγράμματα διαφοροποίησης που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Κατά πρώτον ένα εργοστάσιο στα σύνορα, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, το οποίο βρίσκεται στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσης αυτή τη στιγμή. Και επίσης το θέμα είναι κατά πόσο θα έχουμε και θαλάσσια μεταφορά με ένα ε, λιμάνι που το 2014 ελπίζουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί. Για την ώρα είμαστε στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματός μας για την ολοκληρώση αυτού του έργου. Επίσης ένα άλλο μεγάλο πρόγραμμα είναι ο αγωγός της Βαλτικής, το Baltic Pipe, διότι έτσι με το διάδρομο βορρά και νότου θα μπορέσουμε να διασυνδέσουμε τις σκανδιναβικές χώρες με την υπόλοιπη Ευρώπη με έναν αγωγό που θα περνά από τον πυθμένα της Βαλτικής. Έτσι θα έχουμε δύο σοβαρές διασυνδέσεις σε συνεργασία με την Ελβετία και την Δημοκρατία της Τσεχίας που θα αρχίσουν να λειτουργούν από φέτος τον Σεπτέμβριο και επίσης θα υπάρχει διασύνδεση και με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Το πρόγραμμα αυτό θα καλύπτει 1,5 δις κυβικά μέτρα. Έπειτα, θέλουμε να εξαλείψουμε όλες τις, όλα τα σημεία συμφόρησης που, υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεταξύ της δικής μας αγοράς και της Σλοβακίας, της Λιθουανίας και της, ε, ε, Λιθουανίας προκειμένου να προχωρήσουμε. Έχουμε εκπονήσει σχετικά μελέτη αντικτύπου και μετά την ολοκλήρωσή της θα περάσουμε σε συγκεκριμένες δράσεις. Οι υποδομές αυτές της κεντρικής Ευρώπης, όπως ανανεώνονται, θα αλλάξουν ένα μέρος της αγοράς για την κεντρική Ευρώπη. Όλα όσα κάνουμε, τα πράττουμε έχοντας κατά νου τις γειτονικές μας χώρες και τους εταίρους μας. Έτσι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη αγορά για τη μεταφορά του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Το βασικό μας σχέδιο διαφοροποίησης θα μπορούσε να είναι ένας σταθμός επεξεργασίας του υγροποιημένου αερίου το οποίο λειτουργεί με τρόπο διαφανή, ώστε να υπάρχει πρόσβαση για όλου του εταίρους που θα ήθελαν στο μέλλον να εκμεταλλευτούν αυτή την εγκατάσταση, να, χρησιμο... να ε, συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία υγροποίηση. Διασύνδεση λοιπόν και με τι χώρε τη Βαλτικής, τη Πολωνίας με τις χώρες της Βαλτικής, αλλά και με χώρε τη νότια Ευρώπη, προκειμένου να αναπτυχθούν υποδομέ που να σταματήσουν τι σχέσει εξάρτηση και τα σημεία συμφόρηση στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι θα αναπτυχθεί ο λεγόμενος διάδρομος βορρά-νότου. Και θα δημιουργηθεί ένας νέος αγωγός που θα επιτρέψει την ταχύτερη αξιοποίηση των υπάρχοντων συστημάτων, την ενίσχυση των δικών μας ε, εγχώριων ενεργειακών δικτύων και την αξιοποίηση των υπαρχόντων ευρωπαϊκών. Αυτό στο μέλλον θα μας δώσει δυνατότητες πρόσθετες. Όπως για παράδειγμα, ελπίζω ότι η χρήση του μελλοντικού αγωγού, του Ναμπούκο, θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες ανταγωνιστικότητας και περιορισμό των τιμών του φυσικού αερίου και για τους ε, ιδιώτες, τους καταναλωτές ε, που είναι μεμονωμένοι χρήστες, αλλά και για συλλογικότερα σχέδια. Επίσης υπάρχουν και άλλες προοπτικές. Όπω η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου που ήδη υπάρχει σε κοιτάσματα, στην Πολωνία λόγω χάρη. Θα έρθω κατευθείαν στα συμπεράσματα γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Αυτή είναι η άποψη για συγκεκριμένε θετικέ δράσει στα πλαίσια του προγράμματο προκειμένου να δοθούν κάποιε απαντήσει σε όλα αυτά τα θέματα. Ε, περιμένουμε και τη δική σα ενισφορά, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, και στο μέλλον θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε του περιορισμού στην παροχή φυσικού αερίου χωρίς να ξεχνάμε ότι τα προβλήματα των ενεργειακών συστημάτων πρέπει να αντιμετωπιστούν. Στην ενεργειακή αγορά πρέπει να αξιοποιήσουμε περισσότερο τα διάφορα πλεονεκτήματα που διαθέτει κάθε μεμονωμένη χώρα και να φροντίσουμε να τροφοδοτήσουμε με επενδύσεις τον τομέα αυτό. Οι επενδύσεις βέβαια αυτές, αυτές είναι ιδιαίτερα δαπανηρές, αλλά είναι και χρονοβόρες. Θα πρέπει λοιπόν βράχει πρόθεσμα να δούμε τι δράσεις μπορούμε να αναλάβουμε προκειμένου να πραγματοποιήσουμε μακρόπνοα σχέδια και να έχουμε και μεσοπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα. Για την ενεργειακή μας λοιπόν αγορά θα πρέπει να γίνει μια επιλογή προγραμμάτων τα οποία να στηριχθούν. Οι μηχανισμοί της αγοράς δεν μπορούν μόνοι τους να στηρίξουν τα προγράμματα. Εδώ θέλουμε ε, ολοκλήρωση των συστημάτων τον οποίο μπορούμε να, να μην τον οποίο μπορεί να μην μπορούμε να διαδούμε απευθεία το άμεσο οικονομικό όφελο, όμω θα υπάρξει μεσοπρόθεσμα τέτοιο κέρδο. Επίση υπάρχουν μηχανισμοί που ξεπερνούν την απλή χρηματοδότηση. Μηχανισμοί που έχουν περισσότερο να κάνουν με το κόστος και την απλούστευση την ρυθμιστική, την ε, διοικητική. Χρειάζεται οι διαδικασίες να απλοποιηθούν, ώστε ένα πρόγραμμα να μπορεί σκόπιμα να ετοιμαστεί μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Διότι με όλες αυτές τις διοικητικές καθυστερήσεις τα προγράμματα ετοιμάζονται καθυστερημένα. Αυτό εμποδίζει την πρόθεση της διαφυροποίησης στην Ευρώπη την οποία όμως αν καταφέρουμε να την ε, πραγματοποιήσουμε θα έχουμε μια ενισχυμένη αγορά στην Ευρώπη και να καλύψουμε τις ανάγκες των καταναλωτών. Ε, κλείνω εδώ λέγοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει η περιοχή που όλοι ονειρευόμαστε για την ασφάλεια της παροχής σε φυσικό αέριο και την ενέργεια γενικότερα και εδώ οπωσδήποτε σήμερα λειτουργούμε προσπαθώντας να, να πραγματοποιήσουμε αυτή την ολοκληρωμένη, την ενιαία αγορά φυσικού αερίου. Με τη δική σας στήριξη και συμπαράσταση, με τις καλές σας ιδέες και την ε, θετική σα ενισφορά θα μπορέσουμε να έχουμε τις κατάλληλους μηχανισμούς νομοθετικούς και ρυθμιστικούς. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα ε, στο δεύτερο πάνελ. Ε, θα ακούσουμε τώρα όλες τις ε, ομιλίες για να συζητήσουμε μετά. Στο τέλος θα γίνουν Στο δεύτερο πάνελ θα ασχοληθούμε με το θέμα της τεχνικής και νομικής και της χρηματοδοτικής εφαρμογής. Θα ασχοληθούμε λιγάκι με διαφορετικά θέματα και καλέσαμε τρεις εμπειρογνώμονες, τους οποίους χαιρετίζω θερμά Πρώτος ο κύριος Γκέρλτ Κέντνερ, Αμπριον ε, ε, Transportnets από τη Γερμανία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την δυνατότητα να σας παρουσιάσω τη δική μας άποψη. Εγώ είμαι ασχόλιος για τη διαχείριση κεφαλαίων ε, που περιλαμβάνει και το grid και την εξουσιοδότηση. Μέχρι τώρα είχαμε ε, εξουσιοδότηση για την αναβάθμιση συστημάτων και τώρα αυτά που θα σας παρουσιάσω βασίζονται στην εμπειρία μας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου στο ε, θέμα της ε, αδειοδότησης και να σας αναφέρω ορισμένα πρακτικής φύσεως προβλήματα αλλά και κάποιες λύσεις μπορούν να υπάρξουν. η διαδικασία αδειοδότησης στην Ευρώπη ποικίλει και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί το νομοθετικό πλαίσιο είναι παρεμφερές όπως παραδείγματος χάρη οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτές είναι λίγο πολύ ίδιες σε όλες τις χώρες όμως η εφαρμογή ποικίλει στις διάφορες χώρες και θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα για να οριστεί ε, το σημείο το διασυνοριακό το σημείο επαφής όπως παραδείγματος χάρη ανάμεσα στη Γερμανία Γερμανία και την Ολλανδία, το σημείο αυτό καθορίζεται στο τέλος ε, της εθνικής διαδρομής. Όμως στη Γερμανία ε, το σημείο επαφής είναι το σημείο έναρξη, εκεί που αρχίζει το πρόγραμμα. Βλέπετε λοιπόν ότι ε, δεν μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό. Και επειδή οι διαδικασίες των διαφόρων χωρών δεν συνδέονται μεταξύ τους, πολλές φορές χάνουμε χρόνο και σημειώνονται και καθυστερήσεις. Η δική μας λοιπόν η πρόταση που μπορεί να ε, εφαρμοστεί στην νομοθεσία είναι πρώτα απ' όλα η εναρμόνιση των διαδικασιών αδειοδότησης, κυρίως ε, για όσοι μετέχουν στο δίκτυο. Ένα άλλο θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα ε, κυρίως στους διαδρόμους όπου εφαρμόζονται αυτά τα προγράμματα. Τώρα λοιπόν είναι σχεδόν αδύνατο να βρει κανείς σε κάποιο σημείο που να μην προστατεύεται. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε τη δυνατότητα να μπαίνουμε και ε, σε προστατευμένες περιοχές. Κατά την άποψή μας αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις διαδικασίες στην, ε, ε, στο πλαίσιο της αδειοδότησης. Βέβαια όλοι ξέρετε ότι οι διαδικασίες αυτές είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και ας δούμε τι μπορεί να γίνει. Ε, μέχρι τώρα λοιπόν ε, είχαμε αρκετές ε, χώρες που είχαν διάφορες διαδικασίες αδειοδότησης που ήταν πολύ χρονοβόρες και αυτό που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ θα ήταν να επιτρέψουμε μια απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης οποτεδήποτε χρησιμοποιούνται οι υπάρχοντες ε, διάδρομοι. Ε, ε, το να χρησιμοποιήσει κανείς αυτούς τους διαδρόμους, αυτό θα οδηγούσε στο να αυξηθεί σημαντικά η ισχύ του συστήματος. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το εξής. Έχουμε ε, και επιστημον προδιαγραφές υγείας επιστημονικά τεκμηριωμένες το χάνει για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ε, το 99 μας έκανε συστάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτές πρέπει να επιβεβαιωθούν κατά την άποψή μας. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν μόνο επιστημονικά τεκμηριωμένα όρια. Και εδώ ε, θέλω να αναφέρω και κάτι άλλο. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι να αλλάξει το σύστημά μας σε σύστημα χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα. Βέβαια, οι ε, γραμμές κατασκευάζονται τοπικά και πολλοί ε, αντιδρούν. Ε, βλέπετε λοιπόν πολλές φορές τα τοπικής φύσης προβλήματα πρέπει να ληφθούν και αυτά υπόψη και όχι μόνο τα διεθνή. Και επειδή υπάρχουν τα τοπικής φύσης προβλήματα πολλές φορές δεν επιλύονται τα προβλήματα. Εδώ λοιπόν μιλάμε και για την επικοινωνία. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι πάρα πολλοί άμεσα ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μόνο όταν περνάει ο αγωγός μέσα από την αυλή τους. Και αυτό πια είναι πολύ αργά. Θα πρέπει ε, λοιπόν να υπάρχει σωστή επικοινωνία, είναι παράγοντας επιτυχίας αυτός. Ε, χρειαζόμαστε ε, μια κοινή εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών που πρέπει να στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, τα κρατημέλη, τις εθνικές κυβερνήσεις, κυβερνήσεις κρατηδίων και τους πολιτικούς των κρατών μελών. Αν δεν συνεργαστούν όλοι προς μία κατεύθυνση, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε τη λύση. Έτσι λοιπόν, ε, οι εθνικοί διάδρομοι πρέπει να ανακοινώνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις. Όμως, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ε, είναι σημαντικό να αρχίζει η έγκαιρη ενημέρωση όπως έκανε η εταιρεία μας ε, και όταν το κάναμε αυτό είχαμε πολύ σημαντικές ε, αντιδράσεις. Αυτό είναι στοιχείο κλειδί ε, για να ε, εγκρίνονται οι νέοι αγωγοί. Αυτές λοιπόν είναι οι προτάσεις που είχαμε να κάνουμε για την αδειοδότηση ε, και τώρα θα περάσω σε θέματα χρηματοδότησης. Φέτος είναι γνωστό οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλάζοντας το μέλλον όλο το σκηνικό του ενεργειακού. Αυτό πρέπει να γίνει με προσεκτό κόστος και αξιοπιστία με την έννοια ότι τα συστήματα πρέπει να είναι αξιόπιστα αλλά και η χρηματοδότηση. Η δική μας δουλειά είναι να κατασκευάσουμε και να λειτουργούμε τα δίκτυα ε, να χρεώνουμε τους πελάτες για να προσβέσουμε το κόστος μας και πρέπει να προσελκύσουμε και επενδυτές. Γιατί όπως σας έδειξα και προηγουμένως οι επενδύσεις που χρειάζονται είναι ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε μια αυξανόμενη ζήτηση, ε, για ε, αγωγούς μεγάλων αποστάσεων και αυτό απαιτεί όλο και περισσότερα κονδύλια. Από την άλλη το κεφάλαιο είναι ιδιαίτερα ευέλικτο. Ε, οι επενδυτές δουλεύουν σε παγκόσμιο επίπεδο και βλέπουμε ότι αν οι επενδύσεις είναι ενδιαφέρουσες, είναι μάλλον είναι ενδιαφέρουσες και από πλευράς απόδοσης και από πλευράς κινδύνου. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε ε, ικανοποιητικά κέρδη ε, και χρειαζόμαστε σταθερά επενδυτικά προγράμματα. Εμείς ε, είμαστε εταιρεία που ελέγχεται από ρυθμιστικές αρχές. Ο ρυθμιστής μας είναι και η μεγαλύτερη ευκαιρία μας και ο μεγαλύτερος μας κίνδυνος. Πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Για να ανακεφαλώσω λοιπόν και στο θέμα της ε, χρηματοδότησης, χρειαζόμαστε ικανοποιητικά έσοδα ε, που να είναι αποδεκτά για τις ε, κεφαλαγορές, για τις χρηματαγορές ανά τον κόσμο. Βεβαίως είναι μια πολύ καλή ιδέα το να χρεώνεται η επέκταση δικτύου όπως γίνεται σε αρκετές χώρες του κόσμου. Και επιπλέον πέρα από τα ικανοποιητικά έσοδα πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο. Πολύ σημαντικό αυτό. Και θα ήθελα να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Προηγουμένως αναφέρθηκε ότι ε, για να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα χρειάζονται 10 χρόνια. Εμείς έχουμε κάνει την εμπειρία ότι πράγματι αυτά τα δέκα χρονιά ίσως είναι απαραίτητα ε, και αν αρχίσουμε τώρα την εφαρμογή του προγράμματος δεν θα ξέρουμε το 2020 ε, τι θα έχει προκύψει. Θα έχουμε δηλαδή ίσως τότε άλλους κινδύνους και αν δεν υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο και αν υπάρχει ο κίνδυνος μετά από δέκα χρόνια να πούνε οι αρμόδιες αρχές δεν είναι ικανοποιητικό το πρόγραμμα τότε δεν μπορούμε και να ζητάμε επενδύσεις. Χρειαζόμαστε ένα σταθερό επενδυτικό κλίμα ικανοποιητικά ανταποδοτικά έσοδα και αυτά θα προσελκύσουν τους ε, επενδυτές. Ε, πρέπει λοιπόν να υπάρχει κεφάλαιο χαμηλού κόστους. Ε, αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να αρχίσουν να εφαρμόζονται προγράμματα, αλλά κατά την άποψή μας αυτό δεν είναι ένα πλαίσιο διαρκείας. Για μας αυτό που παίζει ρόλο είναι να υπάρχουν ικανοποιητικά έσοδα και σταθερό πλαίσιο. Αυτά βοηθούν τις επενδύσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ανακεφαλαιώσω όλα τα σημεία που ανέφερα ε, με βάση την πρακτική μας εμπειρία. Χρειαζόμαστε λοιπόν ικανοποιητικά έσοδα για να προσελκύσουμε επενδυτές. Χρειαζόμαστε ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό που μας απασχολεί περισσότερο είναι να επεκταθεί το δίκτυο. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον έχουμε την αμέριστη υποστήριξη όλων των επιπέδων, από επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι και ε, το επίπεδο της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης. Ε, μια μεγάλη βοήθεια θα ήταν να έχουμε απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης σε υπάρχοντες διαδρόμους και επιπλέον αυτό που θα ενδιαφέρει να επιταχυντούν οι διαδικασίες αδειοδότησης. Ευχαριστούμε πολύ λέει ο Πρόεδρος και Επόμενος ομιλητής ο κύριος Ίλαμ Κόλομ ε, που είναι καθηγητής ε, στο Πανεπιστήμιο της ε, Σαραγκόζα στην Ισπανία φυσικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση για να συζητήσω για ένα ευαίσθητο θέμα για την αδειοδότηση υποδομών ε, ε, μεταφοράς ενέργειας. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στην παρέμβασή μου στις διαδικασίες αδειοδότησης αυτής της κατηγορίας υποδομών και θα διαρθρώσω την ε, παρέμβασή μου σε τρία σημεία. Πρώτον, να δούμε ποιος είναι ο στόχος αυτών των διαδικασιών αδοδότησης και τι ακριβώς επισέρχεται. Ένα δεύτερο σημείο θα είναι η υποδομή της διαδικασίας αδειοδότηση και το τρίτο θα αφορά τις ε, αποζημιώσεις που πρέπει να δίνονται στις περιοχές και στους ανθρώπους που δεν ε, ε, λαμβάνουν ε, απευθείας ωφέλη από τα ωφέλη που προέρχονται από τη δημιουργία αυτών των υποδομών. Στο πρώτο σημείο θα ήθελα να επισημάνω ένας, ε, μια δέσμη νομοθετικών ε, ε, μέσων τα οποία προτάθηκαν και μας ενδιαφέρουν για την δημιουργία των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών ενέργειας και έλαβαν υπόψη τους πολύ σημαντικές συνιστώσεις για την επιλογή των έργων τα οποία έχουν σχεδιαστεί. Και αυτό αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προτεραιότητες στις υποδομές. Ξεκινώντας από αυτό το εφαλτήριο, προσπαθήσαμε να δούμε πώς αυτό το νομοθετικό πακέτο που εγκρίθηκε το 2009 είναι επαρκές και να δούμε κατά πόσον θα πρέπει να συμπληρώσουμε κάποια σημεία. Στο πρώτο σημείο της παρέμβασή μας, ε, ο στόχος και το τι υπησέρχεται στη διαδικασία διοδότησης και πιο συγκεκριμένα ξεκινώντας από τη διαδικασία αδειοδότησης αυτή καθεαυτή θα πρέπει να καθορίσουμε τι στόχο έχουμε. Θέλουμε να έχουμε διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς ενέργειας. Θα πρέπει να καθορίσουμε επακριβώς τι εγκαταστάσεις θεωρούμε ότι είναι ε, διευρωπαϊκά δίκτυα ε, χρησιμοποιώντας μια σειρά από τεχνικά κριτήρια τα οποία θα μας επιτρέψουν να γνωρίζουμε τι υποδομές είναι ήδη κατασκευασμένες και είναι και εν εξελίξη και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποτελούν τμήμα αυτών των διευρωπαϊκών δικτύων. Ο λόγος για τον οποίο αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο στόχος αυτό των διαδικασιών αδειοδότηση είναι γιατί απαντούμε στο ε, στο γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ δύσκολο να βρούμε ποια είναι αυτά τα διευρωπαϊκά δίκτυα, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ε, προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όλα αυτά φυσικά εφαρμόζοντας την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 της συνθήκης η αρχή της επικουρικότητας που το 2009 μας οδήγησε ήδη στην έγκριση τριών κανονισμών, των 713, 714 και 715 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις διάφορες πτυχές αυτών των κοινοτικών δικτύων και των φορέων που ε, υπησέρχονται σε αυτά τα δίκτυα. Οι σκέψεις λοιπόν που κάνουμε για τον διευρωπαϊκό χαρακτήρα είναι ε, επικεντρωμένες στο ποιος παρεμβαίνει σε, στα δίκτυα αυτά. Θα παρέμβουν κάποιοι φορές οι οποίοι αναφέρονται στο νομοθετικό πλαίσιο, παραδείγματος χάρη ο Acer, το διαβρικό δίκτυο μεταφορών, οι περιφερειακές ε, αρχές και επίσης θα υπάρχουν και ε, εθνικοί φοροί. Ε, η διαδικασία διαδότησης θα πρέπει να γίνει σε συντονισμένο τρόπο με τους ε, παράγοντες ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τον, τους εθνικούς παράγοντες. Θα περάσω τώρα στο δεύτερο σημείο που αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης. Η διαδικασία διοδότησης θα πρέπει να πληρεί κάποιους βασικούς στόχους, στόχο της διαφάνειας, ε, τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων και επίσης να τηρείται και η αρχή της επικουρικότητας. Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους στόχους, ε, η περίπλοκη διαδικασία της αδειοδότησης θα πρέπει να διαρθρωθεί σε δύο στάδια. Ένα πρώτο στάδιο σε κοινοτικό επίπεδο, στο οποίο στάδιο θα καθορίσουμε τα διάφορα έργα υποδομών ε, σε διαμεθοριακό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη και τον ενεργειακό σχεδιασμό διευρωπαϊκών δικτύων. Και ένα δεύτερο στάδιο, το οποίο θα είναι σε αποκεντρωμένη μορφή και θα πρέπει να αφορά την εκτέλεση του καθενός από τα έργα τα οποία έχουμε καθορίσει προηγουμένως. Και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει συντονισμό μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων σε αυτή την περίπτωση. Η ισχύουσα νομοθεσία αυτή τη στιγμή μας δείχνει την ε, ε, η ευθύνη πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφορών και η νομοθεσία που εγκρίθηκε το 2009 σημαίνει ότι ξεκινάει και μια διαδικασία διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφορώμενα μέρη. Ε, συμμετέχει και η Acer και επίσης λαμβάνεται υπόψη και το περιβάλλον. Αυτός ο σχεδιασμός, ο οποίος ε, είναι στο πρώτο στάδιο, είναι ένας ευέλικτος σχεδιασμός, ο οποίος συντονίζεται με τα εθνικά σχέδια και είναι και συμβατός και με ένα σχεδιασμό σε δεύτερο επίπεδο, σε περιφερειακό ε, πλαίσιο. Ο, το πρώτο αυτό στάδιο είναι πολύ σημαντικό ε, και πολύ καθορισμένο. Θέλουμε να καθορίσουμε τι μας επιτρέπει να έχουμε ένα συνοκτικό δίκαιο μεταφοράς ενέργειας. Στο δεύτερο στάδιο θα περάσουμε στην εφαρμογή του κάθε ενός από τα έργα αυτά. Και εδώ φυσικά μπορεί να υπάρχει και η ανάγκη ανάπτυξης της διαδικασίας για να μπορέσουμε να συντονίσουμε την δράση των κοινοτικών και εθνικών φορέων και επίσης για να αποφύγουμε καθυστερήσεις στην εκτέλεση αυτών των έργων που έχει συζητηθεί ήδη σήμερα το απόγευμα σε πολλές περιπτώσεις. Η νομοθεσία που εγκρίθηκε από το 2009 προβλέπει ότι η ευθύνη είναι των κρατών μελών. Και μόνο το νομοθετικό πακέτο από το 2009 μας επιτρέπει να λάβουμε υπόψη και κάποιους ευρωπαϊκούς φορείς εκ των υστέρων όταν υπάρχουν προσκόμματα στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή θα πρέπει ίσως να τεθεί ε, σε ένα διαφορετικό πλαίσιο και να δούμε κατά πόσον θα ήταν ανάγκη να γίνει συντονισμός εξ αρχής ε, στο δεύτερο στάδιο. Ιδίω όταν αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι να διευκολύνουμε την εκτέλεση των έργων. Και αυτό θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε δίνοντας την ευθύνη στη διαδικασία διοδότησης σε κοινοτικούς φορείς και ε, αυτή η ευθύνη δεν θα απαγόρευε σε κάθε κράτος μέλος να είναι αρμόδιο για το τμήμα της υποδομής που θα αναπτυχθεί εντός της επικράτειάς του. Και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου για το συγκεκριμένο τμήμα του προγράμματο υποδομή. Και φυσικά στο κράτο μέλο θα εκπονηθεί και η πρόταση η οποία θα πρέπει να εγκριθεί υποχρεωτικώ από τον κοινοτικό φορέα, εκτό και αν υπάρχει κάποιο ε, διαφορετικό στόχο, ε, στόχο ο οποίο θα είναι αντίθετο ε, στην πρόταση, στου κοινοτικού κανόνε ή που θα δημιουργούσε πρόβλημα στην, στον ισχύοντα σχεδιασμό και θα ήταν και ε, προβληματικό σε σχέση με άλλο τμήμα της υποδομής που είναι ε, ε, τμήμα άλλης χώρας μέλος. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει μια ενιαία θηρίδα για τις ανακοινώσεις για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την εκτέλεση όλων αυτών των έργων. Όσον αφορά τώρα τις ευθύνες σε αυτούς τους κοινοτικούς φορείς, αυτό θα μας επέτρεπε εξ αρχής να διαπιστώσουμε κατά πόσον υπάρχουν προσκόμματα, να διαπιστώσουμε κατά πόσο υπάρχουν καθυστερήσεις ε, κατά την υλοποίηση του έργου. Επίσης, εάν μπορέσουμε να διευκολύνουμε τις διαδικασίες αδειοδότησης, θα πρέπει ε, να προχωρήσουμε τη διαδικασία αδειοδότησης και να συμπεριλάβουμε και άλλα ε, ίσονο σημασία στοιχεία, όπως για παράδειγμα την ε, άδεια ε, για χρήση γης ή κάποιες άλλες ε, επιπλέον άδειες που θα μπορούσαν να δοθούν και θα είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της υποδομής. Και τελευταίο κομμάτι της παρέμβασής μου, οι αποζομιώσεις στις περιοχές οι οποίες στις οποίες κατασκευάζονται υποδομές. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ποιοι επηρεάζονται από αυτές τις υποδομές και δεν έχουν απευθείας όφελος από το σκοπό των υποδομών και θα πρέπει να τους δοθεί κάποια αποζημίωση. Και αυτή η αποζημίωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα προγράμματα υποδομών, στα οικονομι... στις οικονομικές δαπάνες, για να λάβουμε υπόψη και τις αποζημιώσεις. Οι αποζημιώσεις εννοείται ότι θα πρέπει να είναι και λογικές. Εδώ θα ολοκληρώσω και την παρέμβασή μου για τις διαδικασίες αδειοδότησης των υποδομών ε, μεταφορών ενέργειας σε διευρωπαϊκό επίπεδο και σας ευχαριστώ εκ νέου για την πρόσκληση να συμμετάσχω εδώ σε αυτό το δεύτερο πάνελ που είναι ε, αφιερωμένο στους αδειοδοτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και τώρα ο κύριος Φρανσουά Κλειπό για την δική του παρουσία. Σειρά σας. Σας ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων είναι ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε εδώ και πολλά χρόνια το 87 με 27 κράτη-μέλη. Στόχος είναι να χρηματοδοτεί πολιτικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ενέργεια έχουμε στόχο από τον Οκτώβριο του 2006 για την αξιολόγηση του EIB με την ε, έρευνα στην ενέργεια, την ε, αξιολόγηση της ενεργειακής ασφάλειας και το Διευρωπαϊκό Ενεργειακό Δίκτυο. Θα επικεντρώσω την παρουσίασή μου στη χρηματοδότηση του διενεργειακού δικτύου. Μιλάμε για δίκτυο παροχής και μεταφοράς ενέργειας, το δίκτυο φυσικού αερίου και την αποθήκευση αυτού. Κατά την περίοδο από το 2007 ως το 2010, Περάσαμε από τα 2,5 δις στα 2,7. Εδώ η σωρευτική χρηματοδότηση για τα δίκτυα ενέργειας ήταν 18,2 δις που οδήγησε σε ένα σύνολο 83 επιμέρους επενδυτικών δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων σε 23 διαφορετικά κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και 57 δίκτυα διευρωπαϊκά κοινού ενδιαφέροντος. Οι επενδύσεις που από κοινού υποστηρίχθηκαν έφταξαν τα 56 εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει να σημειώσουμε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη που έχει εντοπίσει 4,2 δις για την ενέργεια και τα προγράμματα υψηλής προτεραιότητας είχε ένα αντίκτυπο επιταχυντικό στα προγράμματα αυτά πέρσι. Η τράπεζα ενέκρινε 1,2 δις ευρώ προκειμένου να υποστηριχθούν 10 προγράμματα που τύχαναν στήριξης από το Ταμείο. Εδώ μιλάμε για την πολυαναμενόμενη διασύνδεση Γαλλίας-Ισπανίας, της Ιρλανδίας και του Ισουαλίας, της Φινλανδίας και της Εστονίας και της Μάλτας με την Ιταλία. 2,4 δις σε δάνεια πρόκειται να δοθούν για προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν το σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην Πολωνία και το νότιο διάδρομο αγωγό φυσικού αερίου. Αυτό που μας προσφέρει το, ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρωπαϊκών Επενδύσεων είναι η συνεισφορά του στην ποιότητα, την ασφάλεια της παροχής και τα οικονομικά πλεονεκτήματα της χρηματοδότησής του. Εδώ μας ενδιαφέρει να δούμε κατά πόσον μπορούμε να σεβαστούμε τους ευρωπαϊκούς στόχους, ιδίως ως προς την βιωσιμότητα σε τρεις συγκεκριμένους τομείς, τον οικονομικό, τον περιβαλλοντικό και τον δημοσιονομικό. Σε ό,τι αφορά το τρίτο σκέλος, Ένα μέρος της χρηματοδότησης ε, τα τελευταία τετραετία είχε να κάνει με συγκεκριμένα μακροπρόθεσμα δάνεια οριμότητας για τους παροχής και υπεύθυνους μεταφοράς ενέργειας που δρούν περιφερειακώς με τους τρεις πυλώνες που μέσα στην τράπεζα έπρεπε πάντοτε να συγκεντρώσουμε με συγκεκριμένους όρους τα κονδύλια προκειμένου να μεταφερθούν στον πελάτη μας με ένα μικρό περιθώριο για να καλύψουν το λειτουργικό τους κόστος. Βέβαια κάποια προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν από συγκεκριμένη δημοσιονομική δομή όπως το εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στην Πολωνία που δημιουργήθηκε από συγκεκριμένη εταιρεία. Let's move now on, on, the future investment need and challenges. Να επικεντρωθούμε τώρα στις μελλοντικές επενδυτικές ανάγκες και τις προκλήσεις μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι για να καλύψουμε το στόχο για το κλίμα και την ενέργεια μέχρι το 2020 χρειάζονται επενδύσεις στα ενεργειακά δίκτυα. 200 δις για τα μεταφορά ενέργειας. Η αξία των επενδύσεων αυτών για την ηλεκτρική ενέργεια είναι ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές και να ενοποιήσουμε τα κυκλώματα. Στον τομέα του αερίου ο βασικός όγκος θα επικεντρωθεί στην διαφοροποίηση και την ασφάλεια της παροχής και σε αυτό σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων επαιτήσεων. Εδώ μας απασχολεί η υπόγεια αποθήκευση του αερίου, η μεταφορά και η βασική αγωγή Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες για αυτές τις επενδύσεις. Πρώτα απ' όλα οι διαδικασίες έναρξης, έπειτα τα θέματα της ρύθμισης, η τιμολογική διάρθρωση, και η σταδιακή επένδυση καθώς και η συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν σχεδιαστεί πάντοτε για να λειτουργούν ανάλογα με την αλλαγή στο επίπεδο των επενδύσεων όπως προβλέπεται για το 2013. Τέλος, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης η πρόσβαση και το κόστος της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης έχουν υποβαθμιστεί. Λίγες παρατηρήσεις για τη δικασία διοδότησης από την εμπειρία μας τα τελευταία χρόνια Και παρόλο που η αδειοδότηση προκαλεί καθυστερήσει για την εκτέλεση των προγραμμάτων, προγραμμάτων έχουν σημειωθεί πρόοδοι. Ήδη του τελευταίου μήνε άρχισε να ισχύει νομοθεσία που προβλέπει αλλαγέ για να ευθυγραμμιστούν οι διαδικασίε. Η στρατηγική και περιβαλλοντική αξιολόγηση, όπως απαιτείται από το άρθρο 142, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να διευκολύνουμε την πρόσληψη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο των νέων υποδομών. Εδώ χρειάζονται και μέτρα αντιστάθμισης και εξισωτικά για να δούμε πώς ε, κάποιες απώλειες θα μπορούμε να τις εξορροπήσουμε για το σχέδιο διασύνδεσης των πόλεων. me I mean, Εδώ λοιπόν πραγματικά είναι επιτακτική ανάγκη να επιταχύνουμε τις επενδύσεις στα έξυπνα δίκτυα. Ενώ σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα συνεχίσει να παρέχει την ε, καλύτερη δυνατή στήριξη για την βιωσιμότητα των προγραμμάτων που αφορούν την διανομή και μεταφορά των ενεργειών με μακροπρόθεσμα δάνεια σύμφωνα με τον οικονομικό κύκλο ζωής των ενεργειακών δικτύων. Αυτή η βασική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα συμπληρωθεί από καινοτόμα εργαλεία που τα μελετούμε αυτή τη στιγμή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρώτα απ' όλα η πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά ομόλογα για την Ευρώπη το 2020. που εγκαινίασαν το Φεβρουάριο ο Επίτροπος Ρεν και ο Πρόεδρος Μαεστάτ, έπειτα να εξεύρουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση για να ενισχύσουμε το πρόγραμμα αυτό των ομολόγων τα οποία θα εκδώσει η αρμόδια εταιρεία και να υπάρξει συντονισμό με το πρόγραμμα που ξεκίνησε πέρσι για να υπάρχει απαραίτητη χρηματοδότηση για την ιεράρχηση των προγραμμάτων υποδομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έπειτα η διευκόλυνση για την χρηματοδότηση των ερευνών, οπότε να διευκολύνουμε τα έξυπνα δίκτυα ή την αποθήκευση ενέργειας και τις σχετικές δράσεις. Πάρα πολύ. Ζαλιστήκαμε από τις πληροφορίες ε, και θέλω να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες ε, που ήταν τόσο σύντομοι και ακριβείς. Ε, αυτό βοηθάει πάρα πολύ γιατί σήμερα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Θέλω όμως να δώσω τη δυνατότητα στους συναδέλφους να υποβάλουν ερωτήσεις. Δέκα έχουν ζητήσει το λόγο και κλείνω ο κατάλογος. Και κατά δεύτερον, όποιος υποβάλλει μία ερώτηση, κοιτάξτε, ε, δεν χρειάζεται να τους ευχαριστείτε εδώ τους ε, συναδέλφους. Τους ευχαρίστησα ήδη. Είναι ευχαριστημένοι. Μετά, να υποβάλουμε ως το δυνατόν περισσότερες ε, ερωτήσεις, γιατί πολλοί εμπειρογνώμονες μπορούν να απαντήσουν μόνο μία ερώτηση και γι' αυτό ε, θα έλεγα ε, ένα έως δύο λεπτά η ερώτηση. Δεν είναι εύκολο, αλλά την συζήτηση μπορούμε να την κάνουμε και μεταξύ μας. Ευχαριστούμε πολύ για την κατανοησία. Η κυρία Ντεκαστήγιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή είμαι η πρώτη, θα ευχαριστήσω εγώ τα μέλη του, μάλλον, ε, του πάνελ και έτσι εκπροσωπώ όλου του συναδέλφου. Δεν χρειάζεται να τους ξαναευχαριστήσει άλλος. Η ερώτησή μου είναι πολύ συγκεκριμένη και θέλω να τη θέσω στον κύριο Ευστάλδιου νομίζω. Μας μίλησε για τα έξυπνα δίχτυα στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ανάπτυξη αυτών των έξυπνων δικτύων πηγαίνει χέρι-χέρι με την ανάπτυξη των υποδομών και των προτεραιοτήτων που έχουμε σε θέματα υποδομών. Σε γενικές γραμμές δεν δίνεται ιδέουσα προσοχή όταν συζητάμε στα θέματα αυτά των υποδομών ε, στα ε, έξυπνα δίκτυα και ορισμένες φορές η προσοχή μας είναι ακόμα λιγότερη από αυτή που δίνεται στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από πλευράς ανάπτυξης πιλωτικών προγραμμάτων επαρκούς μεγέθους ώστε να έχουμε και πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να αξιολογήσουμε τη σχέση κόστους ωφελίας και να μπορέσουμε να αποφασίσουμε όταν θα αναπτυχθούν αυτά τα έξυπνα δίκτυα που έχει μεταξύ άλλων και πολύ ψηλό κόστος αλλά είναι εξίσου απαραίτητα με τις υποδομές μεταφοράς ενέργειας, διότι αλλιώς θα μεταφέρουμε την ενέργεια, αλλά όταν θα πρέπει να ενσωματώσουμε για παράδειγμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή το ηλεκτρονικά οχήματα ή μια αποδοτική κατανάλωση ενέργειας δεν θα υπάρχουν μηχανισμοί εάν δεν αναπτυχθούν καταλήλως και αυτά τα έξυπνα δίκτυα. και επομένως στην Ευρώπη η ανάπτυξη ε, μεγάλων προγραμμάτων, πιλωτικών προγραμμάτων είναι πολύ περίπλοκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί χρειάζονται και επενδύσει και εδώ χρειάζεται και μια κάποια συνεργασία δημόσιου ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων. Σε τι στάδιο βρισκόμασταν λοιπόν την ανάπτυξη έξυπνων ώστε να γίνει η ανάπτυξη με αυστηρό τρόπο και να μην είμαστε μόνο σε θεωρητικό πλαίσιο. Ο κύριος Βέμπερ. Μια ερώτηση προς τον ε, κύριο Ικαρτρός, ο οποίος μας μίλησε για να ανανεώσουμε πηγές ενέργειας. Εσείς δίνετε μεγάλη ελπίδα στην ανάπτυξη αυτών των ε, πηγών ενέργειας για να επιτύχετε και τους ε, στόχους ε, για το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ανοιχτός χώρος σε οικονομικό πλαίσιο και οι κακές γλώσσες πηγαίνουν πολύ πιο πέρα από αυτό που σας λέω εγώ τώρα. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε πολύ ε, ισχυρό ανταγωνισμό από ασιατικές χώρες, κυρίως από την Κίνα, η οποία επενδύει ε, τεράστια ποσά στη χρηματοδότηση αυτών των ε, οικολογικών πηγών ενέργειας, φωτοβολταϊκά και ούτω καθεξής. ουσιαστικά εφαρμόζουν όλες τις μορφές dumping, ε, χρηματοϊκό dumping, ε, υπάρχουν πάρα πολλές επενδύσεις, οι εξαγωγές ε, είναι ούτως ή άλλως με επιδέτηση και αυτό φυσικά έχει σοβαρές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και ο τομέας στην Ευρώπη πλήττεται και αρχίζει σιγά σιγά να εξαφανίζεται διαρωτώ με τι πρέπει να κάνουμε για να ε, προστατεύσουμε αυτές τις επιχειρήσεις του μέλλοντος για να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Oh, ε, ε, ναι, Ο κύριος Μπραζίνα. Συγγνώμη, δεν σας είδα. Δεν, δεν προχωρήσατε γρήγορα, κυρία Φορμπραντ. Η κυρία Φαν Μπραντ και εγώ κρύφτηκα πίσω από το συνάδελφό μου, συμβαίνει καμιά φορά αυτό. Λοιπόν, σύντομα πρόεδρε, βεβαίω ακούσαμε πάρα πολλού ομιλητέ οι οποίοι μα έδωσαν πολλές και ενδιαφέρουσε πληροφορίε. Αυτό όμω που, που έλειψε σήμερα είναι η επίγουσα μορφή. Πιστεύω ότι η υποδομή ενέργειας είναι κάτι ιδιαίτερα επίγον, άρα δηλαδή ε, δεν πρέπει ε, να περιζόμαστε μόνο στην Ιαπωνία, αλλά και στις ανατολικές χώρες ε, έχουμε εξελίξεις. Βλέπουμε πόσο πολύ εξαρτούμεθα από την ενέργεια. Και όσον αφορά την Ευρώπη, εγώ πιστεύω ότι τα σούπερ δίκτυα και τα έξυπνα δίκτυα είναι και τα δύο απόλυτη προτεραιότητα και πρέπει να επεκταθούν ε, κατά τα μέσο, μέσω σε επόμενα έτη. Μία ερώτηση. Πρόκειται για τα έξυπνα δίκτυα. Εκεί έχουν ήδη αναφερθεί αρκετά. Αυτό που μου λείπει είναι η ε, κατάσταση ως έχει τώρα. Ποια είναι τα εμπόδια έτσι ώστε να υλοποιηθούν αυτά τα έξυπνα δίκτυα. Αυτό οφείλεται στην τοπική ε, αυτοδιοίκηση ή ε, εδώ μπορούν να παίξουν ρόλο η εδω μπορεί να παιξουν ρολο η κομισιον και το Κοινοβούλιο. Δεύτερον, ε, αυτά που είπε ο κύριος Τρόστερ σε σχέση με τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας χωρίς υποδομή και προσαρμογή της υποδομής ενέργειας θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ε, υιοθετήσουμε ως προτεραιότητα τις ανώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό όμως δεν γίνεται. Μπορείτε να μας πείτε πού βρίσκονται τα προσκόμματα. Γιατί δεν υπάρχει προτεραιότητα σε αυτά τα δίκτυα. Τι είδου εμπόδια υπάρχουν και τι πρέπει να κάνουμε εμείς ε, βραχυπρόθεσμα ως Ευρώπη. Μπαζιλίνα. Ευχαριστώ θα πρέπει να αναπτύξουμε τις προτεραιότητές μας, όπως είπαμε, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αυτό μας αφήνει μόνο μία εναλλακτική λύση. Αυτό είναι να υπάρχουν ενεργειακοί διάδρομοι, να συνδέσουν τη Βόρεια Ευρώπη και τις ενεργειακές της πηγές με την ε, Νότια Ευρώπη. Και θα πρέπει να υπάρχουν και ευέλικτες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες θα προσθέσουν στα όσα ε, έχουμε αν σταματήσει για παράδειγμα ο άνεμος να φυσάει, ο ήλιος να λάμπει και ούτω καθεξής. Χρειαζόμαστε λοιπόν έξυπνα δίκτυα και υποδομές οι οποίες θα μας επιτρέψουν και να διασυνδεθούμε αλλά και να αποθηκεύουμε την ενέργεια και να τη χρησιμοποιούμε με ευφυή τρόπο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, υπάρχουν παραδοσιακές ε, πηγές ενέργειας ε, οι οποίες θα πρέπει να διασυνδέονται όμως περισσότερο που σημαίνει ότι θα χρειαστούμε περισσότερες επενδύσεις και εδώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι πόροι που θα καταναλώνονται σε τοπικό επίπεδο χωρίς να χρειάζεται να δώσουμε πλέον πόρους για τη μεταφορά της ενέργειας. Και η ερώτησή μου είναι η Έχει εκτιμήσει κάποιος το κόστος εάν όντως αυξηθεί το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχει κάνει κάποιο σύγκριση μεταξύ του κόστους ε, ανανεώσιμων πηγών και παραδοσιακών πηγών ενέργειας. Αν όχι, νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνουμε γιατί το οφείλουμε στον Ευρωπαίο καταναλωτή. Αυτός είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει το κόστος και θα ήθελα να γίνει μια συγκριτική μελέτη. Ο κύριος Κάριντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μία ερώτηση και ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Ε, σήμερα ε, πολλοί από τους ομιλητές είπαν ότι είναι απαραίτητο να ενταχθούν, να ενσωματωθούν οι ανώσιμες πηγές ενέργειας και τα έξυπνα δίκτυα. Και άλλοι μίλησαν για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Κανείς όμως δεν μίλησε για το ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει κοινή αγορά και θεωρώ ότι το έκανε γιατί όλοι θεωρούν ότι είναι δεδομένο, όχι ότι δεν τους ενδιαφέρει για να αυξηθεί η χρήση ε, των ανώσιμων πηγών ενέργειας ε, πρέπει να αυξήσουμε τα έξυπνα δίκτυα. Όμως για την ασφάλεια του εφοδιασμού ε, και για την περίπτωση τη δυνατότητα να υλοποιηθεί μια αγορά χρειαζόμαστε τις γραμμές διασύνδεσης. Και εδώ έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Τρέστερ Στην ομιλία σας ε, αυτό που ήταν πολύ ενδιαφέρον ήταν όταν μιλήσατε για το σούπερ δίκτυο ε, τον βορειοαφρικανικό ήλιο ή το τόξο αυτό φαντάζομαι της Βορειοαφρικής. Αν μπορούμε να συνδυάσουμε τον ήλιο της Βόρειας Αφρικής ε, και τον ε, άνεμο της Βόρειας Θάλασσας θα έχουμε θαυμάσια αποτελέσματα. Ε, στη Βαλτική, παραδείγματος χάρη, αυτό μπορείτε να δείτε και στη διαφάνεια, η Βαλτική όλη η περιοχή της Βαλτικής είναι εκτός της Ευρώπης στην παρουσίασή σας. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το εξετάσουμε. Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρουσίαση ήταν της της κυρίας Τσιρλίτσοβα. Εσείς ε, εκπροσωπείτε 33 εταιρείε και 22 χώρες και καμία από αυτές δεν είναι από τις χώρες της Βαλτικής γιατί το ε, Gazprom ε, που έχει το μονοπόλιο όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται, αλλά είναι και παντελώ αποκομμένη η Gazprom από την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν από αυτές τις συζητήσει που είναι πολύ ενδιαφέρουσες, ε, θέλω να πω το εξή. Αν πραγματικά μας ενδιαφέρει η ενιαία αγορά και το super δίκτυο και η ασφάλεια μου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη βορειοανατολικά τη Ευρώπη υπάρχει ένα ενεργειακό νησί, ε, το οποίο για πάρα πολλούς λόγους ε, πρέπει και αυτό να ενταχθεί ε, στο ε, δίκτυο. Η κυρία ε, Φαρέρα Μαντουρέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να περάσω απευθεία στο προκείμενο, στον κύριο Καρβάγιο. Εσείς είπατε πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε την ενέργεια που παράγεται στη Βόρεια Αφρική και να την ε, περάσουμε στην ε, Ευρώπη και αναφερθήκατε και σε ένα διάδρομο νοτιοανατολικό. Μήπως θα έπρεπε να έχουμε και έναν ε, διάδρομο βορρά-νότου, όπως γίνεται με το φυσικό αέριο και όχι μόνο για τον νοτιοανατολικό διάδρομο. Επίσης, αναφερθήκατε στα δεκαετή προγράμματα ανάπτυξης και είπατε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό όραμα. Τι θα πρέπει να κάνουμε για το ευρωπαϊκό αυτό όραμα, τι ιδέες έχετε εσείς. Και τέλος, την κυρία Τσιρλίκοβα. Θα ήθελα να γνωρίζω σε τι φορά και σε ποιες πλατφόρμες θα συζητηθούν τα θέματα αυτά και θα δούμε ποια προγράμματα θεωρούνται προτεραιότητα. Υπάρχει κάποιος ρόλος, μπορούν να πούν κάτι οι ομάδες ε, περιφερειακών πρωτοβουλειών ή θα δημιουργηθούν συγκεκριμένες ομάδες και συγκεκριμένες πλατφόρμες για να συζητήσουν αυτό το ζήτημα. Ο κύριος Κύριος Γκλάντε, ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση και μία παρατήρηση. Ο συνάδελφος μου ρώτησε ε, σε ποιο επίπεδο πρέπει να γίνει κάτι. Νομίζω και στα δύο επίπεδα, και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να το χάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν θα υπάρχουν προτεραιότητες ε, για τους αγωγούς, ε, θα πρέπει κανείς να διερωτηθεί τι πρέπει να υπερισχύει, η αγωγή ή η χλωρίδα και η πανίδα. Γι' αυτό πρέπει να συζητηθεί, το θέμα αυτό πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, σε εθνικό επίπεδο ε, και μιλάω έχοντας κατά νου τη δική μου περιφέρεια, έχω πάρα πολλά παραδείγματα ε, για το κατά πόσον το αέριο είναι εναλλακτική ενέργεια. Ε, δεν υπάρχει σχεδόν κανένας τομέας όπου να μην ασκείται πίεση από πλευράς πολιτών. Προηγουμένως ο κύριος Κένελ έθιξε ένα άλλο θέμα ε, σχετικά με τη ε, διαδικασία διαδότησης και την επιτάχυνσή της. Νομίζω ότι ε, το να υπάρξει περιορισμός σύντμηση της διαδικασίας αυτής, αυτό δεν νομίζω ότι γίνεται. Οι άλλες διαδικασίες πρέπει να περιστούν είναι πιο αποτελεσματικές, έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να κατατεθούν ε, πολλές αριθμητικά εφέσεις. Εμείς ε, ε, έχουμε στην Γερμανία κάποιες πρωτοβουλίες, εκεί οι πολίτες δεν συμμετέχουν. Όταν όμως φτάνει ο γερανός, τότε ενδιαφέρονται όλοι. Αυτό που ενδιαφέρει επίσης είναι το πώς είναι δυνατόν να γίνει, ε, να γίνει ανανέωση δικτύων. Σε μένα, ας πούμε, οι πολίτες ε, είπαν ε, να παραμείνουν εγωγοί, απλά να εξυγχρονιστούν. Εσείς τι λέτε, βοηθάει αυτό και έχετε εμπειρία από αυτού. Η κυρία Τίκαου. Που δεν είναι εδώ, θα έρθει λίγο ο κύριος Οντί. Ευχαριστώ, Ήθελα να σας πω ποια είναι η προσωπική μου εντύπωση. Όταν ακούω όλους τους προσκεκλημένους μας που όλοι έχουν ιδιαίτερα προσόντα, με ε, αφήνει άφωνο το πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα στην Ευρώπη. Και το θέμα είναι και ποιος έχει την κατοχή των δικτύων. Ποιος έχει την κατοχή του τα δίκτυα. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι μια μέρα δεν θα καταλήξουμε σε πλήρη αταξία ως προς το, την ιδιοκτησία. Α υποθέσουμε ότι την Γκάσπρομ αγοράζει ένα δίκτυο αύριο, του το απαγορεύει, της το απαγορεύει η νομοθεσία, άραγε υπάρχει για το τι λειτουργήσε και τι όχι στα διάφορα κάτι μέλη σε σχέση με την εγκατάσταση των δικτύων οδικών, σιδηροδρομικών, και ούτω καθεξής. Για να υπάρχει δηλαδή μια πολιτική ευρωπαϊκή Διερωτώ με, δεν θα έπρεπε να έχουμε μια τελικά υπερετερία κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θηγατρική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που να έχει στα χέρια της τη διαχείριση των δικτύων και να καθορίζει τις τιμές για τους καταναλωτές διότι δεν μπορώ να σκεφτώ σε τι μπορεί να εξυπηρετήσει τους καταναλωτές όλη αυτή η περιπλοκότητα και για την ηλεκτρική ενέργεια και για τον αέριο. Ο κύριος Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούσαμε πολλά στοιχεία που δεν γνωρίζαμε σήμερα. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τους συναδέλφους ιδιαίτερο τον κύριο Κάρινς, που έκανε λόγο για νησίδες ενέργειας ή για στήριξη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι το σύστημα ενέργειας δεν είναι νέο στην Ευρώπη και ότι θα πρέπει να το στηρίξουμε. Στην Βαλτική Ένωση θέλουμε να συμπαρασταθούμε στις προσπάθειες αυτές για συμπερίληψη του όλου δικτύου τους στο ευρωπαϊκό σύστημα. Χρειάζεται όμως και ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός. Σήμερα εξεπλάγει από κάποιες αναφορές. Όταν μιλάμε για ηλεκτρικό δυναμικό. Φαίνεται να μην είμαστε ακόμη έτοιμοι να διαχειριστούμε την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Προσπαθούμε να μεταρρυθμίσουμε διάφορες πολιτικές που βλέπουμε όμως στην πράξη να μην λειτουργούν. Τρία θεσμικά όργανα τρεις θεσμοί ευρωπαϊκοί θα έπρεπε να διαθετούν τις βασικότερες αρχές που έχουν να κάνουν με τον τομέα του φυσικού αερίου. Και αυτοί οι τρεις θεσμοί δεν έχουν κοινή προσέγγιση μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα από τα βασικά εμπόδια που μας δυσκολεύει. Επίσης, κανείς δεν έκανε λόγο σύστημα σήμερα για την αντιστροφή του συστήματος. Ένα σύστημα που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την παροχή αερίου. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο σύστημα. Πρέπει να δημιουργηθεί άμεσα μέσα στην ερχόμενη διετία. Πρέπει να τοθεί το ζήτημα του συστήματος αυτού, διότι αν δεν λειτουργήσει άμεσα, τα ανατολικά κράτη δεν θα μπορέσουν ποτέ να διασυνδεθούν με το δικτικό δίκτυο. Κοιτάξτε, εγώ προτείνω ε, το εξής θα σας δώσω σε όλους τη δυνατότητα ε, να απαντήσετε εφόσον το επιθυμείτε και αν κάποιος ε, θεωρεί από τους ομιλητές ε, ότι δεν τον αφορά κάποια ερώτηση μπορούμε να, μπορεί να περάσει επόμενος. Ο κύριος Ροζίτης καταρχήν. Ναι. Μου θέσετε μία ερώτηση για το 18 πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου και είπατε ότι δεν είναι και τόσο ευρωπαϊκό το όραμα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το δεκαετές πρόγραμμα και γίνεται στα πλαίσια της ανάπτυξης που προβλέπεται ε, σε κάθε κράτος μέλος. Είναι ένα σύνολο όλων αυτών και κάθε κράτος μέλος κάνει το σχεδιασμά του και μετά έγινε μία σύνοψη και συμπεριέλαβε όλα τα ε, προγράμματα που προγραμματίζονται. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό όραμα, αν θέλετε, διότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε χώρα όταν αναπτύσσει το δίκτυό της οδηγούν Ε, στο εξή φαινόμενο. Πολλές χώρες ε, είναι πολύ λιγότερο επιθετικέ από όσο θα έπρεπε για την ανάπτυξη των δικτύων τους και σε κάποιες χώρες αυτό μπορεί να εξαρτάται και να ε, δυσχεραίνεται από συγκεκριμένες ε, εξελίξεις και έργα τα οποία θα πρέπει να γίνουν για να είναι θετικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο ελπίζω για την επόμενη διαδικασία αυτών των προγραμμάτων των δεκαετών να καθοριστούν κάποια αρχικά κριτήρια τα οποία θα προκύψουν από τα όσα γνωρίζει πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάθε κράτος μέλος θα κάνει το σχεδιασμό του από εκεί και πέρα. Ο σχεδιασμός όμως θα πρέπει στη συνέχεια να συντονιστεί ή να ενδυναμωθεί από τις υπόλοιπες χώρες ώστε να επιτύχουμε αυτό το ευρωπαϊκό όραμα το οποίο θα πρέπει να υπάρχει μέσα σε αυτά τα δεκαετή προγράμματα. Ευχαριστώ. Ε, if you want. Ο κύριος Ελφστάντιους. Καταρχήν, ε, όσον αφορά την ερώτηση σχετικά με τα, ε, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δίκτυα διανομής κατά το παρελθόν όταν επρόκειτο να υπάρξει νέα τεχνολογία, ετίθεται το θέμα της ε, συνεργασίας ανάμεσα στους οργανισμούς κοινής ωφελία και τους ε, ε, παρόχους ε, τεχνολογίας. Κατά το παρελθόν η συνεργασία ήταν σε διμερές επίπεδο. Τώρα όμως, όταν μιλάμε για έξυπνα δίκτυα, και αν δούμε λιγάκι την κατάσταση ε, σε επίπεδο διανομής όπου ε, συμπεριλαμβάνεται και ο χρήστης, ε, ξαφνικά έχουμε πάρα πολλούς άμεσα ενδιαφερόμενους. Έχουμε τους καταναλωτές, Έχουμε τις εταιρείε κατασκευής, τους παρόχους επικοινωνίας, τους παρόχους εξοπλισμού, τον χειριστή του δικτύου και άλλες ε, πιο παραδοσιακές μορφές ε, παροχής ενέργειας. Για να συντονιστούν λοιπόν όλα αυτά, ε, αυτό που ενδιαφέρει είναι τα εμπορικά κίνητρα, τα επιχειρηματικά μοντέλα, όπου πρέπει να καθορίσουμε ένα πλαίσιο συνεργασία λοιπόν με τις αρχές και που μεγάλο ρόλο παίζουν και οι πολιτικές. Γι' αυτό για μας η έρευνα και η ανάπτυξη είναι πολύ σημαντικό ε, για να αναπτυχθούν, για να αντιμετωπίσουν τα σωστά, σωστά τα θέματα. Και συμφωνώ ότι ίσως υπάρχουν χώρες ε, που είναι πιο προχωρημένες, αλλά πιστεύω ότι στην Ευρώπη έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες ε, για να αναλάβουμε τα ενία αυτών των εξελίξεων. Και νομίζω ότι εδώ οι κυβερνήσεις ε, πρέπει να εξετάσουν το θέμα. Και όσον αφορά τώρα ε, το στοιχείο αν είναι τοπικό ή όχι. Ε, πράγματι πρέπει να δούμε και ξέρουμε ότι υπάρχει εθνικό πλαίσιο αλλά υπάρχει και κοινοτικό πλαίσιο. Και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει διάλογος σε τοπικό αλλά και σε ε, κοινοτικό επίπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε λοιπόν να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή αγορά που θα στηρίζει το έξυπνο δίκτυο γιατί μιλάμε για ενεργούς ε, καταναλωτές και μιλάμε και για μια αγορά που, που, που καθοδηγείται από τον καταναλωτή. Αυτή είναι η όλη ιδέα του έξυπνου δικτύου. Ο κύριος Τρούστα. Ευχαριστώ ετέθησαν κάποια ερωτήματα ε, και ελπίζω να τα σημείωσα καλά. Νομίζω λοιπόν το πρώτο ερώτημα αφορά ε, το πιλωτικό πρόγραμμα ε, έξυπνο δίκτυο. Στην Δανία έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ με αυτό το πρόγραμμα και το καλοκαίρι θα υπάρξει και δοκιμή σε δίκτυο διανομής. Νομίζω λοιπόν εκεί υπάρχει κάποια κίνηση. Το θέμα είναι κατά πόσο έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε και κάποια σύγκριση ως προς την εξοικονόμηση διοξιδίων του άνθρακα. Το δεύτερο ερώτημα αφορά σε προϊόντα στην προστασία των ανώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη. Αυτό δεν αφορά μόνο τις ανανεώσιμες αφορά και άλλα προϊόντα. Και εγώ δεν είμαι εδώ ειδικό όσον αφορά αυτό το θέμα. Γι' αυτό δεν θέλω να πω τίποτα από αυτού. Όσον αφορά τώρα ε, στα κατεπήγοντα, ε, κατά πόσον είναι επίγον να έχουμε ένα έξυπνο δίκτυο ή ένα σούπερ δίκτυο, εγώ θεωρώ ότι ε, το σούπερ δίκτυο ή η επέκταση του υπάρχοντος δικτύου, κατά την άποψή μου, αυτό θα πρέπει να έχει προτεραιότητα. Γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ε, χρησιμοποιήσουμε μεγάλη ποσότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μεγάλο δίκτυο και ο χρόνος προγραμματισμού είναι και πολύ μεγάλος. Βεβαίως στο μέλλον θα παίξουν τα δίκτυα κάποιο ρόλο. Ακούσαμε ε, το θέμα της ε, ανάπτυξής τους και κατέστησε αφές ότι χρειαζόμαστε ακόμα χρόνο για να φτάσουμε εκεί. Το ερώτημα γιατί οι χώρες της Βαλτικής δεν συμπεριλαμβάνονται πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Εδώ μεταξύ περιλαμβάνονται στο μοντέλο μας. Αλλά τότε δεν είχαμε αρκετές πληροφορίες και το είπα αυτό στην ομιλία μου ότι εμείς σε γενικές γραμμές ενδιαφερόμαστε και έχει νόημα πράγματι ε, να δώσουμε στην δημοσιότητα ε, δεδομένα έτσι ώστε να είναι δυνατόν να διεξαχθούν και οι απαραίτητες μελέτες από μελετητικά γραφεία όπως το δικό μας παραδείγματο χάρη. Ε, εμείς την ολιγορία δεν την είδαμε τόσο τραγική αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα βελτιωθήκαμε. Έτσι κι αυτό έχει να κάνει ε, με την κατανάλωση και εν πάση περιπτώσει τώρα είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι για καλύτερες μελέτες στο μέλλον. Δεν έχω ε, να σας πω τίποτα άλλο. Ε, αυτά είχα να σας πω. Ο κύριος Τασνόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Έχω σημειώσει αρκετέ ερωτήσει, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Καταρχά απελευθέρωση σε σύγκριση με τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια στην απελευθέρωση, ο κύριος στόχος της, ε, των ενεργειακών υποδομών ήταν να δημιουργήσουμε κοινέ αγορές και να απελευθερώσουμε την αγορά. Μετά όμως άρχισε η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, και οι δυνατότητες απελευθέρωσης αγοράς είναι περιορισμένες πλέον, διότι οι δυνατότητές μας μειώνονται. Και ο λόγος είναι ότι έχουμε πλέον ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι δύο ε, πηγές αντιβαίνουν η μία στην άλλη. Δεν χρειαζόμαστε μόνο διασύνδεση, αλλά θα πρέπει να ε, αποφεύγουμε και τις ε, συμφορήσεις στα συστήματα μετάδοσης ενέργειας. Είναι σαν να ε, προσθέτουμε μία τέταρτη λωρίδα σε έναν αυτοκινητόδρομο και μετά ο αυτοκινητόδρομος ε, να συνεχίζει να λειτουργεί ε, με ένα μικρό δρόμο σε ένα άλλο σημείο. Αυτό είναι η συμφόρηση. Και αυτό διαπιστώνουμε. Έγινε μια ερώτηση για την επένδυση στα δίκτυα. Μπορώ να σας δώσω τα αριθμητικά στοιχεία στη Τσεχική Δημοκρατία. Δεν ξέρω τα στοιχεία πανευρωπαϊκά, αλλά αυτή τη στιγμή γίνονται τεράστιες επενδύσεις. Η ευθύνη για την ασφάλεια τώρα. Ποιος είναι υπεύθυνο ε, για την ε, ασφάλεια εφοδιασμού. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια και έχουν διαβιβάσει αυτή την ευθύνη στους διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς. Επομένως, την τελική ευθύνη έχουν οι διαχειριστές συστημάτων, οι TSOs. Δεν θα πρέπει να επενδύουμε λοιπόν μόνο σε ε, μετασχηματιστές, σε γραμμές, σε διαδρόμους, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει μια ισορροπία και η συνολική ευθύνη είναι για τους ε, διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς. Τώρα, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Στην Τσεχική Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 1.700 ε, ΜΒ σε ηλιακούς συλλέκτες. Τα περισσότερα οι περισσότεροι από αυτούς τους ηλιακούς συλλέκτες προέρχονται από την Κίνα. Επομένως, ε, κάποια τεχνολογικά επιτεύγματα είναι αδιανόητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ε, τα χρησιμοποιούμε, αλλά δεν, τα αγοράσαμε από άλλους και αυτό σημαίνει ότι τεχνολογικώς δεν εξελισσόμεθα. Uh, Ευχαριστώ. Δέκα λεπτά είναι πολύ λίγος χρόνος για να αναπτύξει καλής όλα τα περίπλοκα σημεία Σε ό,τι αφορά την συμπερίληψη των κρατών της Βαλτικής, είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή κανένας από τους ε, επόπτες των συστημάτων, τους διαχειριστές των συστημάτων ε, δεν έχει υποβάλει αίτηση για να γίνει παρατηρητής. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι διαχειριστές των κρατών της Βαλτικής δεν είχαν καμία συμμετοχή στα προγράμματα. Συμμετείχαν και στην περίοδο του 2011-2013 και τα συστήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν και για τις δοκιμές αντοχή του Ευρωπαϊκού Συστήματος, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φυσικού Αερίου, προκειμένου να ενσωματωθούν στα πορίσματα της διαδικασίας αξιολόγησης για την αντοχή. Θα τα βρείτε αυτά στις επιπλέον διαφάνειες που σας έχω μοιράσει. Uh, τα προβλήματα της Βαλτικής πρέπει να αντιμετωπιστούν επιγόντως και να δούμε τι γίνεται με τα περιφερειακά δίκτυα παραγωγής ενέργειας. Ε, um, Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με τις ε, διάφορες περιφέρειες. Και το 2015 να δούμε ποια γραμμή προτείνεται και από τα συμπεράσματα του, του Συμβουλίου. Ως προς το φόρουμ που αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα και ενδιαφέροντα, δεν ξέρουμε ποια είναι τα κριτήρια για αυτά τα προγράμματα. Ας δούμε ποια είναι τα φόρουμ που πρέπει να συζητήσουν τα βασικά προγράμματα και ποια θα είναι τα... ποιες θα είναι οι διαστάσεις των προγραμμάτων αυτών. Τη συγκεκριμένη χρονιά Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα φόρα που ήδη προβλέπονται για την περιφερειακή συνεργασία. Καθώς και τα ήδη υπάρχοντα επενδυτικά προγράμματα. Για την ανάπτυξη λοιπόν τέτοιων προγραμμάτων θα φροντίσουμε να χρησιμοποιήσουμε την πλέον αποτελεσματική διαδικασία για να ενισχύσουμε τους πόρους των ε, διαχειριστών κατά τον ε, πλέον κατάλληλο τρόπο. Ο στόχος δεν είναι μόνο οι υποδομές αλλά και άλλα στοιχεία που πρέπει να αξιοποιήσουν οι διαχειριστές. TSO. Και μια απάντηση στην ερώτηση για το ποιος έχει την ιδιοκτησία των δικτύων. Δύσκολο να απαντηθεί αυτό Δύσκολο να καθησυχήσουμε τις ανησυχίες. Ίσως η διαδικασία απλούστευσης που προλεπτωθεί το ενεργειακό πακέτο να διευκολύνει τα πράγματα. Ο κύριος Τσέλαμ. Bardzo krótko, tylko w kontekście tego ostatniego pytania, które zostało zadane dotyczące likwidacji wysp i działań. Κοιτάξτε, όσον αφορά την ερώτηση που έγινε σχετικά ε, με την ε, ε, κατάργηση και την μία αναφορά των ε, νησιών. Εγώ είπα ότι πρέπει να έχουμε μία πιο αυστηρή πολιτική ενσωμάτωσης. Ακριβώς για να μπορούμε να διασφαλίσουμε τη διασύνδεση ανάμεσα στα δίκτυα. Και εδώ μάλιστα πρότεινα και κάτι και κατόπιν επανέλαβα τις ε, προσπάθειες που γίνονται σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς υπάρχουν ε, ακόμα και χρηματοδοτικά κίνητρα τα οποία επιτρέπουν να ολοκληρωθεί ε, η αγορά. Η επιτυχία εξαρτάται κυρίως από τη συνεργασία σε επίπεδο φορέων εκμετάλλευσης, ε, σε επίπεδο κρατών μελών και κατόπιν χρειάζεται και χρειάζεται και ε, όθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, που να αφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και άλλους φορείς. Ευχαριστώ πολύ. Κατά πρώτον, να δούμε τα πράγματα στη σωστή τους προοπτική. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι απαραίτητα μια μικρή περιορισμένη πηγή. Μπορεί να είναι μεγάλη εμβέλεια η παραγωγή αυτή. Σκεφτείτε ας πούμε τι γίνεται με τις εγκαταστάσεις για αιωλική ενέργεια υπερακτίως. Εδώ έχουμε σκεφτεί πως μπορούμε στα έξυπνα δίκτυα να συμπεριλάβουμε και αυτές τις μορφές. Και για τα έξυπνα δίκτυα η μεταφορά που προβλέπετε είναι ήδη έξυπνη εφής, αλλά το θέμα είναι τα έξυπνα δίκτυα από την άποψη της διανομής, όχι της μεταφοράς. Εκεί χρειάζεται περισσότερο δυναμικό. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έδισα ίσω αρκετή έμφαση στην παρουσίασή μου. Το χρειαζόμαστε αυτό και μάλιστα σύντομα. Γι' αυτό για την ερώτηση του κυρίου Γκλάντε, για το πώ θα επιταχύνουμε τι διαδικασίε μα. αυτό θα ήθελα να επισημάνω. Επίση, χρειαζόμαστε καλή επικοινωνιακή πολιτική. Επικοινωνιακή πολιτική και από την Ευρωπαϊκή Ένωση έω το επίπεδο των ε, αρχών τοπική αυτοδιοίκηση. Χρειαζόμαστε σταθερούς νόμους, σταθερό νομοθετικό πλαίσιο στη Γερμανία. Άλλαξαν πολλές φορές σχετικοί νόμοι τα τελευταία χρόνια, γιατί υπήρξαν και πολιτικές ε, αλλαγέ. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι αυτό μπορεί να οδηγεί σε έλλειψη ασφάλειας. Το σταθερό νομοθετικό πλαίσιο είναι καθοριστικής σημασία. Απλώ μια μικρή λεπτομέρεια εδώ. Χρειαζόμαστε και κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες ε, θέσεις των αρχών και με τα απαραίτητα κονδύλια στη διάθεσή τους. Τριπλασιάσαμε τον αριθμό των εργαζομένων ε, που χειρίζονται τα προγράμματα και τις διαδικασίες, όμως από την ε, πλευρά των αρχών μειώθηκαν ε, οι εργαζόμενοι. Άρα δεν μπορούν να διαχειριστούν τα προγράμματα. Εδώ να επιμείνω ότι οι αρχές είναι εκείνες που διαβάζουν τα προγράμματα δεν θα πρέπει όμω να εμπλέκονται σε τέτοιε διαδικασίε σε προεκλογική περίοδο. Για τη χρήση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων και υποδομών έχουμε την παραγωγή των 720 κιλοβάτ. Αυτή, των 220 κιλοβάτ έχουμε αυτή τη δυνατότητα το να χρησιμοποιούμε τις απαραίτητες γραμμές παραγωγής είναι πολύ αποτελεσματικό. Έχει αποδειχθεί αυτό επανειλημμένος. Και επίσης απέχουμε μόνο ένα βήμα από την νομοθεσία έτσι όπως προβλέπετε με το δικαστήριο που θα αποφασίσει τελικά. Μόνο ένα μπορεί να αποφασίσει. Κύριε Τρεβό. Έγιναν κάποιες ερωτήσεις για τη Βαλτική και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Uh, Baltic Energy Market Integration Plan is a key element. Uh, Το βασικό σχέδιο αυτό ολοκλήρωση είναι ένα απόσπαστο στοιχείο τη ολοκλήρωση του ενεργειακού δικτύου που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ε, απλώ ε, περιλαμβάνει τι ανανεώσιμε περιοχέ, αλλά μα ενδιαφέρει και η βαλτική περιοχή. Έχει γίνει κάποια πρόοδος στον ε, τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχει μια νέα γραμμή μεταξύ Φιλανδίας και Εστονίας, η οποία προχωράει. Υπάρχει και μια νέα γραμμή μεταξύ Σουηδίας και Λιθουανίας. Στον τομέα του φυσικού αερίου ε, θα καθυστερήσουμε λίγο περισσότερο, αλλά υπάρχει ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Πολωνία που μπορεί να θεωρηθεί το πρώτο στάδιο και μετά θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με τη Βαλτική. Για τα έξυπνα δίκτυα συμφωνώ απολύτως. Ε, είναι ήδη ε, κάτι το οποίο υπάρχει στο σύστημα ε, μεταφοράς και υπάρχουν και κάποιες επενδύσεις οι οποίες γίνονται σε έξυπνα δίκτυα. Γίνονται πολλές επενδύσεις για να εγκαταστήσουμε ευφύς μετρητές στον τελικό καταναλωτή, στον τελικό χρήστη. Γίνονται λοιπόν παρά τα εμπόδια όλα αυτά. θα πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή σε κοινά πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον εξοπλισμό και αυτό το αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υπάρξει και σχετική πρόταση νομοθεσίας του χρόνου, επομένως θα αρθεί ένα από τα βασικά εμπόδια για περαιτέρω επενδύσεις ε, και όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα. Αν θυμάμαι καλά, τα έξυπνα δίκτυα είναι επιλέξιμα προγράμματα στην πρωτοβουλία η οποία είναι εξελίξει αυτή τη στιγμή για τη διαδικασία διοδότησης τώρα. Έγιναν πολλές ερωτήσεις για το πώς μπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία διοδότησης. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένα συνδυασμός διαφόρων πραγμάτων. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στην εθνική νομοθεσία για να μειωθεί ο αριθμός των αρχών που συμμετέχουν ε, στην ε, διαδικασία διοδότησης και για προγράμματα υψηλής προτεραιότητας ίσως ε, θα πρέπει να περάσουμε σε εθνικό επίπεδο απευθεία. Η κατάλληλη τώρα τη στρατηγική αξιολόγηση αντικτύπου, όπω ανέφερα νωρίτερα, είναι ένα από τα χρήσιμα μέσα για να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς βέβαια θα πρέπει να συνεχίσουν να ενισχύουν τη δυνατότητα τους ε, να ασχολούνται με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και να ε, εισαγάγουν αυτή τη συζήτηση στο ευρύ κοινό και φυσικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ίσως πιο δαπανηρή μεν τεχνολογία, αλλά τεχνολογία η οποία θα μπορεί να επιταχύνει την εφαρμογή κάποιων ε, από αυτά τα προγράμματα. Ε, η εφαρμογή της κόκκινης ε, γραμμής, για παράδειγμα, είναι ένα καλό παράδειγμα. Ο κύριος Καμπαλιοζόζα ήθελε απλώ ε, να προσθέσει μία πρόταση, άντε το πολύ τρεις, λέει ο πρόεδρος. Ναι, αν κατάλαβα καλά, κάποια στιγμή υπήρχε κάποια αντίθεση μεταξύ των έξυπνων δικτύων και των υπερδικτύων. Ε, είναι συμπληρωματικά τα δύο. Τα έξυπνα δίκτυα θα βοηθήσουν περισσότερο τη ζήτηση, ενώ τα υπερδίκτυα θα βοηθήσουν με τη χρήση της, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην πηγή τους. Αυτή τη στιγμή, όπως χρησιμοποιείται το σύστημα σε κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει να προσθεθεί ένα υπερδίκτυο και ένα ευφυές δίκτυο ε, ανάλογα ε, με τη ζήτηση. Ένα από τα θέματα λοιπόν τα οποία θα πρέπει να δούμε είναι πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το συντονισμό των TSOs για να μπορούν να δράσουν μέσω της ολοκλήρωσης αυτής της ενέργειας για να μπορέσουμε να φτάσουμε από την περιφέρεια στο σημείο κατανάλωσης. Επίσης αναφέρθηκε και το θέμα της αγοράς και της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη δυνατότητα διασύνδεσης. το γεγονός ότι είναι ευμετάβλητο το θέμα των ανανεώσιμων πηγών τη ενέργεια και δεν μπορούμε να προβλέψουμε πόσο χρήση θα μπορούμε να κάνουμε, μας δυσχεραίνει ε, στη λύση μας Και επομένως ε, επειδή μπορεί να υπάρξει διασύνδεση, μπορεί να περιορίσει αυτό που μας μείνει για το εμπόριο. Ε, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία λοιπόν μας καταδεικνύουν ότι η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να έχουν επίσης και αυξημένες δυνατότητες ε, διασύνδεσης. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, εμπειρογνώμονες και όλους ε, τους ε, συναδέλφους για το ότι πράγματι στην ώρα μας τελειώσαμε. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Παρ' όλα αυτά νομίζω η ακρόαση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, αποκτήσαμε πολλές πληροφορίες. Και πριν κλείσουμε θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Βάγνα, ο οποίος είχε πολλή δουλειά και θα έχει ακόμα περισσότερη για να κλείσει το όλο θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς, αποδείχθηκε στη σημερινή συνεδρίαση πόσο ενδιαφέρει τις πολιτικές ομάδες ε, και πόσο καλά έκαναν ε, που επέλεξαν αυτούς τους ανθρώπους ε, να έρθουν εδώ για να μας διαφωτίσουν για όλα αυτά τα θέματα. Ακούγοντάς τους να μιλούν, πιστεύω ότι δόξα τω Θεώ ο κανονισμός δεν μας επιτρέπει να κάνουμε μια δεύτερη δημόσια κρέωση εμπειρογνωμόνων γιατί θα ξαναφέρουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι παραπάνω ειδικοί όπως πρέπει, παραπάνω ευθύς από όσο πρέπει και θα μας φορτώσουμε περισσότερα προβλήματα για ένα θέμα το οποίο ούτως ή άλλως από μόνο του έχει πολλά και δύσκολα προβλήματα. Ευχαριστώ λοιπόν όλους όσους ε, μίλησαν, ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες, ευχαριστώ και τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση και εμείς θα συνεχίσουμε. Αύριο το πρωί έχουμε και άλλη συνεδρίαση που θα συζητήσουμε το ίδιο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, uh, please, uh, can I interrupt for some minutes, please? Uh, there will be... Θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση γιατί υπήρξε μια ε, συνέντευξη τύπου για καθυστέρησε η συνέντευξη τύπου. Αυτοί δεν τελείωσαν στην ώρα του, όπω τελείωσαμε εμεί. Να η διαφορά ανάμεσα στην Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Εκείνοι αργούν, εμεί πάντα στην ώρα μα. Βλέπετε. 5-6 λεπτά καθυστέρηση λοιπόν. So, liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir müssen doch noch mal ein bisschen. Ich habe zwar eben gesagt, die sollen bitte dieses Rollo wieder hochmachen, damit wir nicht hier. Κοιτάξτε, ανοίξτε τι κουρτίνε. Δεν μα αρέσει εδώ ε, να καθόμαστε, σαν, ε, είμαστε σε υπόγειο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν αυτοί που έχουν τι ε, κάμερε ε, και ε, τις θέλουν να κατέβουν οι κουρτίνε για να μπορούν να έχουν καλύτερη εικόνα. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει. Εγώ θέλω να δω τον ήλιο, λέει ο πρόεδρο. Ε, μια φορά που έχουμε και ήλιο, ε, να το ευχαριστηθούμε και λιγάκι. Τέλο πάντων, ήρθε και ο επίτροπο ή έρχεται, είναι καθοδόν. Ja, meine Damen und Herren, ich darf äh, Sie alle begrüßen. Nein, die meisten haben wir ja schon gesehen, weil wir ja schon lange Sitzungen hatten und alle anwesend waren. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε σήμερα τόσους πολλούς προσκεκλημένους ε, και ε, χαιρετίζω θερμά τον Επίτροπο κ. Ότιγκερ, ο οποίος ε, θα μας δώσει πληροφορίες για την αξιολόγηση της κατάστασης στην Ιαπωνία πιο συγκεκριμένα των πυρηνικών εργοστασίων στην Ιαπωνία. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μπόρεσε να έρθει αυτήν την εβδομάδα, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν. Και είναι ιδιαίτερα κατάλληλη η χρονική στιγμή σήμερα, γιατί ε, γίνεται και η συζήτηση με τους υπουργού από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έγινε αυτή η συζήτηση και έτσι θα έχουμε και πολύ επίκαιρες πληροφορίες. Βεβαίω, βλέπω όλοι θέλετε να υποβάλλετε ερωτήσεις. Ε, γράφω τα ονόματά σας. Εν πάση ο συνάδελφος κύριος Οίτιγκερ θα κάνει μια μικρή εισαγωγή και μετά θα έρθετε, είναι η σειρά σας, με τις ερωτήσεις που θέλετε να υποβάλλετε. Ε, κύριε Οίτιγκερ, ε, σας δίνω το λόγο. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής. πράγματι, Αυτά που συνέβησαν στην Ιαπωνία οδήγησαν στο να πρέπει να διαβουλευτούμε επιγόντως και σίγουρα υπάρχουν επιπτώσεις στην Ευρώπη. Όσον αφορά τα συναισθήματά μας, θέλω να πω το εξή. Εγώ προσωπικά πριν από μία εβδομάδα δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα έβλεπα στη ζωή μου τέτοιες εικόνες. Και μερικοί από εσά ε, μιλάτε για αποκάλυψη χρησιμοποιείται αυτή τη λέξη, θεωρώ λοιπόν ότι πράγματι πρόκειται ε, για ένα δόκιμο όρο. Αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία επικρατεί ησυχία. Η ώρα εκεί είναι περίπου δύο τη νύχτα. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε και τις τελευταίες ειδήσει. Όμως εγώ ανησυχώ πάρα πολύ και για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Μετά από όλα αυτά που ακούμε σε αυτό το μεγάλο πυρηνικό εργοστάσιο με 4.700 ΜΒ παραγωγή και 6 διαφορετικές υπομονάδες, σχεδόν τα πάντα είναι εκτός ελέγχου. Οι Ιάπωνες και δικαίως θεωρούνται ως ε, ιδιαίτερα ικανοί ε, τεχνο, τεχνικοί, πολύ καλοί εμπειρογνώμονες, ε, γνωρίζουν καλά τα θέματα, σεβόμαστε τα προϊόντα τους και τη δουλειά τους ε, και πολύ σωστά κάνουμε, αλλά... Όσον αφορά την κατάσταση επιτόπου, σας είπα, είναι εκτός ελέγχου. Η ψυχραιμία και γενικά ο έλεγχος μιας τέτοιας ποινική εγκατάστασης έχει χαθεί. Γι' αυτό λοιπόν το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι να μας φυλάξει ο Θεός. Ο Θεός φυλάξει. Ο Θεός φυλάξει αυτές και τις επόμενες ώρες για να μην γίνει τίποτα ακόμα χειρότερο. Κατόπιν τούτου λοιπόν είναι ακόμα σημαντικότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συζητήσουμε για τις ε, συνέπειες. Ε, το κάναμε αυτό στην Κομισιόν τις τελευταίες ημέρες ε, σε επίπεδο ομάδας εργασίας. Ήρθαμε σε επαφή με, την, με τον, την διεθνή, τον Διεθνή Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας στη Βιέννη. Ήρθαμε σε επαφή με το γραφείο μας που μας αντιπροσωπεύει στο Τόκιο. Απευθυνθήκαμε σε όλους που μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες και σήμερα το πρωί είχαμε την πρώτη συνάντηση υψηλού επίπεδου με τα κράτη-μέλη και τους υπουργούς εκπροσώπους. Είχαμε και υπουργούς και ανώτατα στελέχη υπουργείων. Συναντηθήκαμε δηλαδή με όλους όσοι έχουν να κάνουν με την πυρηνική ενέργεια σε επίπεδο κρατών μελών. Συναντηθήκαμε επίσης και με όλες τις ε, επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, φέρουν ευθύνη για κάποια πυρηνικά εργοστάσια και συναντηθήκαμε και με τους ε, παραγωγούς πυρηνικής ενέργειας από τη Γαλλία, από την Ευρώπη και από την Αμερική. Συζητήσαμε διεξοδικά την κατάσταση και το τι μέλη γενέστε. Και πρέπει να σας πω, είμαι ευγνώμων για το ότι ε, όλοι οι μετέχοντες θέλουν να δείξουν την κοινή ευρωπαϊκή στάση, δήλωσαν ότι είναι πρόθυμοι να διεξάγουν έκτακτα τεστ καταπώνησης με στόχο να αναζητηθούν τα κοινά κριτήρια η αναζήτηση ενδεχομένου κινδύνων, ενδεχομένου κινδύνου μετά από όλα αυτά τα οποία έγιναν στην Ιαπωνία. Άρα δηλαδή σήμερα κανείς ε, δεν ε, οχυρώθηκε μόνος του πίσω από στεγανά, αλλά όλοι αποφασίσαμε ότι θα διεξάγουμε, όπως σας είπα, τεστ καταπώνησης, ε, θα δεχτούμε τις γνωμοδοτήσεις ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, θα τους επιλέξουμε όλοι από κοινού. Εκεί λοιπόν δεν τίθεται θέμα κράτους μέλους, γιατί κανείς δεν είχε αρνητική άποψη επ' αυτού. Στη νέα αξιολόγηση των κινδύνων ε, θα τεθεί και το θέμα της, ε, των σεισμών μετά τα δεκτενόμενα ε, στην Ιαπωνία. Επίσης το παλιροϊκό κύμα, το τσουνάμι στον Ατλαντικό που μπορεί να πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις. Θα τεθεί επίση το θέμα των τρομοκρατικών ενεργειών, των ψυκτικών συστημάτων και των εγγύσεων λειτουργίας τους, το θέμα της διακοπής παροχής ενέργειας, το θέμα της ποιότητας και του δυναμικού των έκτακτων συστημάτων παροχής ενέργειας ε, των πυρηνικών εργοστασίων, το θέμα του, της ηλικία ε, του τύπου κατασκευής ε, και του έτους κατασκευής. Υπάρχει μια οδηγία περιπινικής ενέργειας που εγκρίνατε εσείς και που βρίσκεται ενισχύ αυτή τη στιγμή, τον Ιούλιο συγκεκριμένα του 2011, μέχρι τον Ιούλιο θα πρέπει να έχει ε, μεταφραστεί ε, στα κράτη-μέλη, θα πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στην νομοθεσία τους. Μέχρι το 2014 η οδηγία αυτή προβλέπει ότι θα πρέπει ε, να υπάρχει ε, μέχρι τότε και ένας ενδιάμεσος απολογισμός. Εμείς λοιπόν είμαστε αποφασισμένοι αυτόν τον ενδιάμεσο απολογισμό να τον προτάξουμε χρονικά για να δούμε κατά πόσον είναι δυνατόν ε, να επεκτείνουμε τις οδηγίες που υπάρχουν και σε άλλους τομείς μετά από την εφαρμογή των ε, τεστ καταπώνησης έτσι ώστε να ε, καταλήξουμε όπως σας είπα σε συγκεκριμένες ε, διατάξεις σχετικά με την πυρηνική ενέργεια. Εξάλλου, χαίρομαι της υποστήριξης των μετεχόντων στην ομάδα υψηλού επίπεδου οι οποίοι ενέκριναν ε, τα τεστ ε, καταπώνησης όχι μόνο στα 27 κράτη-μέλη αλλά και στις όμορες χώρες όπως ε, στην Ελβετία, στην Τουρκία, τη Ρωσία. Ελέγχθη λοιπόν ότι και εκεί πρέπει να γίνουν οι δοκιμές αυτές γιατί η ασφάλεια δεν σταματάει στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εχθές λοιπόν συναντήθηκα με το Γενικό Διευθυντή ε, ε, του Διεθνούς Οργανισμού Πυρηνικής ε, Ενέργειας, του έστειλα πιο συγκεκριμένα μια επιστολή στη Βιέννη και τον παρακάλεσα εκεί να συζητηθούν οι συνέπειες μετά τα τεκτενόμενα στην Ιαπωνία, να αναζητηθούν, να αναζητηθούν νέες προδιαγραφές και βέβαια ίσως να μην πρέπει ε, να το πω, αλλά παρόλα αυτά θα πω ότι ο κύριος ε, Σαρκοζή ε, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των G20 ως πρόεδρος ε, θα θελήσει να προσθέσει ε, στα θέματα και το θέμα της ε, Ιαπωνίας. Σήμερα συζητήσατε εσείς, αύριο θα συζητήσει και η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου και θεωρώ ότι Δευτέρα θα έχουμε μια έκτακτη σύγκληση του Υπουργείου Ενέργειας παράλληλα και το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που είναι αρμόδιο για την Euratom και έχω και την υποψία ότι ο κύριος Βαν Ρόμπεϊ την επόμενη εβδομάδα ε, στο έκτακτο συμβούλιο δεν θα μιλήσει μόνο για θέματα προεπλογισμού και δημοσιονομικά, αλλά θα αποδώσει ιδιαίτερη σημασία και στο θέμα της Ιαπωνίας. Αυτά είχα να σας πω προς το παρόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα έχω ένα ανεπίλητο, δυσεπίλητο ε, θα έλεγα πρόβλημα και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε σε επίπεδο πολιτικών ομάδων. 26 έχουν ζητήσει το λόγο. Αντικειμενικά αυτό δεν γίνεται γιατί πρέπει να τελειώσουμε στις 6.30 ε, και φαντάζομαι ότι θα θέλετε να έχετε και απάντηση στην ερώτησή σας. Άρα δηλαδή πρέπει να ε, περιστεί δραστικά ο αριθμός των ερωτώντων. Μισό λεπτό, μην ξεκινήσουμε τώρα να τσακωνόμαστε. Ναι, αλλά σύντομα σας παρακαλώ. Εγώ θα πρότεινα ε, καταρχήν από κάθε πολιτική ομάδα ε, να λάβει ένα στο λόγο και μετά θα δείτε. Εντάξει, σύμφωνοι. Λοιπόν, ο κύριος Βιντάλ Κουάντρας έχει το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον ε, κύριο Επίτροπο για την παρουσίασή του η οποία ήταν ήρεμη, αντικειμενική και σοβαρή, όπως ακριβώς ε, αρμόζει σε τέτοιες περιστάσεις. Βρισκόμαστε ενώπιον ενός πολύ σοβαρού πυρηνικού ατυχήματος. Ε, κατά πάσα πιθανότητα θα ε, υπάρξουν πολύ σοβαρά προβλήματα σε ένα πυρηνικό σταθμό 40 ετών. Ένα ατύχημα το οποίο σίγουρα θα έχει συνέπειες οι οποίες θα διαρκέσουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα παρά το γεγονός ότι η γεωγραφική έκταση του ατυχήματος, αντίθετα με αυτό που συνέβη στο Τσερλομπέιλ, θα είναι περιορισμένη σε όλη την ιστορία των σημαντικών ε, πυρηνικών ατυχημάτων όπως το Τζερνομπίλ ε, μάθαμε κάποια μαθήματα και το συγκεκριμένο ατύχημα θα μας ε, μάθει κάποια πράγματα και εσείς ουσιαστικά μας δώσατε και κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε πλήρως. Υπάρχουν δύο προκλήσεις αγαπητοί συνάδελφοι τις οποίες θα πρέπει να αποφύγουμε. Η μία είναι βραχυπρόθεσμη και δεύτερη είναι ο πανικός. Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται υπό την επίδραση συναισθηματικών ε, εντάσεων και ε, κοιτώντας κοντόφθαλμα ε, στο άμεσο μέλλον είναι συνήθως λανθασμένες. Να μην ξεχνάμε το γενικό πλαίσιο του προβλήματός μας της ενέργειας. Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές κατά 80% μέχρι τα μέσα του αιώνα και μέσα σε 50 ή 40 χρόνια η κατανάλωση ενέργειας ενεργειας παγκοσμιως θα έχει πολλαπλασιαστεί ε, Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση η οποία είναι αναπόφευκτη. Και έχουμε μία σειρά από μέσα και δεν θα πρέπει να χάσουμε κανένα από αυτά τα μέσα. Και όπως είπε και ο Επίτροπος, πολύ λογικά θα πρέπει να σκεφτούμε την Ευρώπη. Θα πρέπει να σκεφτούμε τις περιστάσεις και τα χαρακτηριστικά της Ευρώπης. Και σε αυτή την περίπτωση να σκεφτούμε τις φυσικές καταστροφές και να ε, προσανατολιστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό ακριβώς σας περιμένουμε τι θα γίνει, να μάθουμε τι έχουμε να μάθουμε από όλη αυτή τη διαδικασία και όταν θα λάβουμε τις αποφάσεις μας, οι οποίες θα είναι καρπός αυτών ε, που συνέβησαν, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, θα πρέπει να είμαστε ε, διανοητικώς ε, έτοιμοι και πολιτικά υπεύθυνοι. Ευχαριστώ κυρία Εκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο για την παρουσία του εδώ βιώνουμε δραματικές στιγμές και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για το πώς επηρεάζει όλη η κατάσταση την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και πώς θεωρείτε ε, ότι ελήφθησαν οι αποφάσεις για το ε, κάθε ενεργειακό μείγμα της κάθε χώρας και πιστεύω ότι και άλλες χώρες ε, θα λάβουν ανάλογες αποφάσεις με αυτές που ακούσαμε. Η κυρία Χάρμς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Οτίνγκερ που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας. Ε, θα ήθελα, ε, όπως τα έχω ακούσει εγώ τουλάχιστον και όπως τα έχω καταλάβει αυτά περί Ιαπωνίας, να κάνω μια παρατήρηση και παρακαλώ πάρα πολύ να ληφθεί υπόψη στη συζήτησή μας. Στην Ιαπωνία υπήρχε εμπειρία με μεγάλους σεισμούς και με σημαντικές ζημιές σε πυρηνικά εργοστάσια. Νομίζω το 2007 τότε ήμουνα στην Ιαπωνία, το Κασιουβαζάκι, ε, ε, καταστράφηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό έτσι ώστε από τις 8 μονάδες σήμερα μόνο 3 να λειτουργούν και τότε ε, κυρίως ε, η Χιμπακούσα, οι επι, ε, επιζώντες του Ναγκασάκη και της Χιροσίμα είπαν την άποψή τους, εμφανίστηκαν στο προσκήνιο και είπαν ότι η Ιαπωνία, στην Ιαπωνία δεν πρέπει να την ποινική ενέργεια. Αυτό δεν τον είπαν άνθρωποι εκτός Ιαπωνίας, αλλά μέσα στην Ιαπωνία και η προειδοποίηση αυτή με το Κασιμπαζάκι, αυτό τον ε, πυρηνικό σταθμό, προφανώς αγνοήθηκε, να ήταν ληφθεί υπόψη. Και αν σας κατάλαβα καλά, σήμερα βρισκόμαστε όλοι εδώ για να δούμε πώς πρέπει να ερμηνεύουμε τις προειδοποίησεις. Τις τελευταίες ημέρες άκουσα το φίλο σας, τον κύριο Τόπφερ, ο οποίος είπε ότι όταν εκείνος ήταν υπουργό Περιβάλλοντος, ε, κατάλαβε ότι η διαδικασία τήξης σε πυρηνικό εργοστάσιο διεξάγεται ανεξέλεγκτα και είπε ότι για αυτό το λόγο πρέπει να εγκαταλείψει η Γερμανία το στομό των δυνατών την πυρηνική ενέργεια. Εγώ λοιπόν ρωτώ ε, κατά πόσον ακριβώς αυτή η άποψη του κυρίου Τέπφερ που την εκφράζει επιθετικά εδώ και πολλά χρόνια ε, το κατά πόσον ατυχήματα πυρηνικής ε, σε οποιονδήποτε αντιδραστήρα και σε οποιαδήποτε χώρα δεν περιορίζονται στον υποδοχέα ε, ε, θα ήθελα λοιπόν να ξέρω κατά πόσο αυτά που μας λέτε παίζουν, έχουν σχέση με τα τεστ καταπώνησης τα οποία θα διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Τσίτσεστερ, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που ήρθατε εδώ κύριε Επίτροπε. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζουμε μία ταχαίως εναλλασσόμενη κατάσταση. Τα νέα τα οποία έρχονται από την Ιαπωνία ε, είναι από βαθιά αισιοδοξία μέχρι μετριοπαθή, ε, συγγνώμη, από βαθιά αισιοδοξία μέχρι μετριοπαθή αισιοδοξία για το τι συμβαίνει στο ε, πυρηνικό αντιδραστήρα της Φουκουσίμα. Στην Ιαπωνία βιώσαμε μια εξαιρετική φυσική καταστροφή, είχαμε ένα σεισμό και ένα τσουνάμι και θα πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι τι ακριβώς συνέβη πριν αρχίσουμε να κάνουμε παραλληλισμούς με την κατάσταση στην Ευρώπη. Θα ήθελα να υποστηρίξω τον συνάδελφο Βιντάλ Κουάντρα και να πω και εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μην δράσουμε βεβαιασμένα. Έχουμε ήδη κάποια μέτρα, τα έχουμε εφαρμόσει και να είμαστε λίγο πιο καθησυχασμένοι να δούμε τι ακριβώς συνέβη πριν ε, λάβουμε περαιτέρω μέτρα. Να σας υπενθυμίσω αγαπητοί συνάδελφοι ότι η Ευρώπη εξαρτάται από την ε, πυρηνική ενέργεια για το 30% της ηλεκτρικής της παροχής όσοι θέλουν να εξαφανιστεί η πυρηνική ενέργεια ε, και καταφέρουν να περάσει το δικό τους, ε, θα, νιώθουμε, θα βιώσουμε τα προβλήματα διακοπής ενέργειας που βιώνουν αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία, επειδή ακριβώς υπήρχαν προβλήματα στον πυρηνικό σταθμό. Ας είμαστε ψύχρεμοι. Ο κύριος η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Επιτρόπε, που ήρθατε μαζί μας απόψε το απόγευμα να μας εξηγήσετε πώς έχουν τα πράγματα. Νομίζω πρώτα απ' όλα στο όνομα της Επιτροπής Ήτρε, όχι μόνο των σοσιαλιστών αλλά όλων των συναδέλφων, πρέπει να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς την Ιαπωνία και τον Ιαπωνικό λαό. Και επίσης πρέπει να αποτίσουμε φορό τιμής σε όσους εργάζονται σκληρά για να προλάβουν όλες τις απώλειες που μπορεί να προκύψουν από, την, από το πυρηνικό εργοστάσιο στην ε, Ιαπωνία. Να σταθεροποιηθεί η κατάσταση είναι η πρώτη μας μέρημνα. Και για εκείνους και για μας. Είναι πολύ σημαντικό. Έπειτα, νομίζω ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητές μας για να ελέγξουμε τις δικές μας τις ευθύνε. Να δούμε ποιε είναι. Και η πλέον επιτακτική ανάγκη για τους Ευρωπαίους ηγέτες είναι να ενημερωθεί ο ευρωπαϊκό πληθυσμό και να ενημερώνεται διαρκώ για την εξέλιξη της κατάστασης και τον κίνδυνο. Άρα ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προεδρία του Συμβουλίου να εξασφαλίσουν ότι θα συγκεντρώσουν εμπειρογνώμονε για να παρακολουθούν την κατάσταση στενά και να ενημερώνουν διαρκώ το ευρωπαϊκό κοινό. Ε, ο πανικό είναι ο χειρότερο σύμβουλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Προεδρία θα πρέπει να διαπραγματευτούν με, την διεθνή, με το Διεθνή Οργανισμό για την Πυρηνική Ενέργεια καθώ και την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνική ενέργειας και κάθε άλλο ειδικό που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να ε, ξεφύγουμε αλόβητα από αυτή την κατάσταση. Επίσης, άλλη επιτακτική ανάγκη είναι, εφόσον βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να βρούμε έναν τρόπο να βοηθήσουμε την Ιαπωνία, να διορθώσει το πρόβλημα όσο το δυνατόν συντομότερα. Πρέπει λοιπόν να καλέσουμε την Επιτροπή να οργανώσει ανθρωπιστική βοήθεια και επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη όσο το δυνατόν συντομότερα και να αποσταλούν επιτόπου στην Ιαπωνία. Είναι επιτακτική ανάγκη αυτή πρέπει να διασφαλίσουμε όχι μόνο του πολίτε, αλλά και τη στατιωτική και μη στατιωτική χρήση και να εξασφαλίσουμε όλα αυτά τα εργαλεία που διαθέτουμε για τέτοιου είδου παρεμβάσει. Η άλλη ευθύνη μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ευρωπαϊκή. Η ευρωπαϊκή που αφορά τα όσα προκύπτουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε και να βελτιώσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ασφάλεια της πυρηνική ενέργειας σε όλη την Ήπειρο για οποιαδήποτε παραγωγή, οποιοδήποτε είδου. Ε, θα συμφωνήσω εδώ με όσα είπατε και για τι γειτονικέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει αυτό. Και θα πρέπει να επικεντρωθούμε όχι μόνο στην πυρηνική ενέργεια και την ασφάλειά τη, αλλά να θυμίσω στου συναδέλφου και το τι έγινε πριν από ένα μόλι χρόνο άλλου είδους ε, καταστροφή λόγω παραγωγής ενέργειας που πρέπει να την ε, ελέγξουμε. Δεν ε, οφείλεται σε φυσική ε, καταστροφή αλλά σε ανθρωπογενείς παράγοντες. Πρέπει λοιπόν να καθησυχάσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες ότι τις γνώσεις μας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και την ασφάλειά της μπορούμε να τις βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε να παρακολουθούμε το τι συμβαίνει προσεκτικά. Και έπειτα αφού συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες, όλα τα στοιχεία πρέπει να αντλήσουμε τα κατάλληλα διδάγματα για να λάβουμε μακροπρόθεσμε αποφάσει. Συνάδελφοι, θέλω να ολοκληρώσω λέγοντα το εξή για να αποφύγουμε την πολιτική αλυσιδωτή αντίδραση πρέπει να ασκήσουμε τις ευθύνες μας και πρέπει να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα με ε, δραστηριότητε ελέγχου. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Πέτρο που ήρθατε εδώ. Ε, δεν θα επαναλάβω όλους τους άλλους συναδέλφους όσα είπαν. Απλώς πρέπει και εγώ να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Κουάντρα, την κυρία Χέρτσοκ και τον κύριο Τσίτεστερ. Ε, απλώς θέλω να θέσω μία ερώτηση. Οι διαβουλεύσεις θα γίνουν με τη συμμετοχή της Ρωσίας που έχει τέτοιες εμπειρίες καθότι είναι και γειτονική χώρα της Ιαπωνίας. Μίλησαν λοιπόν όλες οι πολιτικές ομάδες ε, και τώρα θα προχωρήσω. Παρακαλώ όμως ε, μόνο ένα λεπτό καθένας για να έχουν την ευκαιρία όσο το δυνατόν ε, περισσότεροι. Επόμενος κυρία Ντελκαστίγιο. Για να μην καθυστερήσουμε πολύ, δεν θα παρέμβω γιατί θεωρώ ότι οι προηγούμενες παρεμβάσεις στην πλειονότητα τους ε, εξέφρασαν και τις δικές μου απόψεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Οντή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων που προλάβατε να έχετε με την Επιτροπή μας. Πρώτα απ' όλα θα χαιρετήσω την τόλμη και την αξιοπρέπεια του Ιαπωνικού λαού για την δοκιμασία που περνάνε. Ε, εδώ πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας διεθνώ και λυπούμε που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προβλέψει την Ευρωπαϊκή Δύναμη Προστασίας των Πολιτών, που θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη σε αυτήν την κατάσταση. Ήδη από το 2010 είχαμε την έκρηξη της πετρελαϊκής πλατφόρμας και αυτό το σοβαρότατο ατύχημα το είχαμε ήδη περάσει. Ε, Ξέρουμε μάλλον ότι δεν μπορούμε να παράγουμε ενέργεια με μηδενικό κίνδυνο. Σήμερα λοιπόν η πολιτική τη Επιτροπή πρέπει να αναθεωρηθεί. Η έρευνα, η ανάπτυξη, ό,τι αφορά την ασφάλεια τη παροχή, οι κλιματικέ αλλαγέ, οι δεσμεύσει μα σε διεθνέ επίπεδο. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Επίση, η πυρηνική ενέργεια εντό κοινότητα, ευρωπαϊκή κοινότητα για την πυρηνική ενέργεια. Θα πρέπει η έρευνα, η ασφάλεια, τα διεθνή πρότυπα που θα μας επιτρέψουν ε, να βελτιώσουμε το επίπεδο προστασίας μας ε, προς το όφελος των Ευρωπαίων πολιτών, να έχουμε καλύτερες προδιαγραφές για αυτή την, του είδους την ενέργεια που όμως είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την παρουσία του και για το γεγονός ότι έδρασε ταχύτατα. Εδώ και αρκετό καιρό θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στραφεί περισσότερο στο μέλλον της ενεργειακής μας πολιτικής και θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι έχουμε προβλήματα ε, αντίστασης. Ε, ναι, θα πρέπει να καθορίσουμε μια σειρά από κριτήρια. Αλλά υπάρχει ένα κριτήριο το οποίο θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αυτό είναι η ημερομηνία κατασκευής ενός πυρηνικού αντιδραστήρα. Στο Βέλγιο αλλά και στη Γαλλία πολλοί από αυτούς τους πυρηνικούς σταθμούς ε, ε χρονολογούνται από τη δεκαετία του 70. Είναι ήδη 40 ετών, έχουμε πάνω από 400 ε, πυρηνικούς σταθμούς και είναι πολύ παλιότεροι από την ε, δεκαετία του 70. Στην Ιαπωνία συνέβη κάτι ασύλληπτο. Δεν έχουμε όμως εμπειρία για τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν αυτοί οι πυρηνικοί ε, αντιδραστήρες που είναι τόσο παλιοί. Εμένα με στεναχωρεί το γεγονός ότι γίνεται επιλεκτική ε, ε, ε στην κατάσταση και δεν κοιτάμε ότι πρέπει να έχουμε ένα νέο ενεργειακό μήκο. Κύριε Πίτροπε, Υπήρχε από ό,τι ακούσαμε συμφωνία να γίνουν κάποια τεστ καταπώνηση για τα περισσότερα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω με ανησυχεί και αυτό, διότι υπάρχει ένα πράγμα που νομίζω ότι δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το προβλέψουμε ήδη από το, όσα συνέβησαν στην Ιαπωνία. Ο σεισμό, αυτό καθεαυτό, δεν ήταν το αίτιο του προβλήματο. Ο σεισμό πυροδότησε την απόφαση να κλείσει το αντιδραστήρα. Ο αντιδραστήρα σταμάτησε να λειτουργεί και μετά προέκυψε το πρόβλημα. Αυτό, η έκρηξη που έγινε μετά δημιούργησε την όλη κατάσταση. Στα τεστ καταπώνησης που γίνονται και ασχολούμαστε με επιμέρους προβλήματα, είναι άλλο αυτό που κάνουμε. Στην Ιαπωνία συνέβη κάτι που θα μπορούσε να συμβεί και στην Ευρώπη χωρίς κανένα σεισμό. Ε, εδώ το θέμα είναι η πολύπλοκη και αλυσιδωτή αυτή καταστροφή όπως έλαβε χώρα. Και αυτό που μας απασχολεί είναι ότι η διαδικασία ασφάλεια με ένα απλό τεστ καταπώνηση δεν βλέπει τι συμβαίνει σφαιρικά. Όταν συμβεί μια τέτοια φυσική καταστροφή, προφανώ βρίσκεται κανεί σε τέτοια θέση όπου η ε, απλή λήψη μέτρων, τα κλασικά μέτρα δεν λειτουργούν πλέον. Είναι πολύ πλοκότερο το σύστημα των προβλημάτων. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν θα έχουμε μια ευρύτερη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Η κυρία Ριμπάζη. Ευχαριστούμε κύριε Έντιγκερ που είστε μαζί μας. Ε, πρέπει να πω ότι μιλήσαμε εδώ για ατύχημα, μετά έγινε λόγος για καταστροφή, για αποκάλυψη. Ε, νομίζω ότι ωραίους χαρακτηρισμούς βρήκαμε για την κατάσταση στην Ιαπωνία, όμως η Ευρώπη έχει σοβαρότατες ευθύνες για την ε, ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας. Όταν δούμε λοιπόν την κατάσταση της Ιαπωνίας, μας υποχρεώνει αυτό να δούμε ξανά το πώς έχουμε αξιολογήσει του κινδύνου. Εκεί συσσωρεύτηκαν πολλοί κίνδυνοι μαζί. Ε, ο σεισμός, το τσουνάμι, το παλαιροϊκό κύμα που πλημμύρισε τα συστήματα αυτά ηλεκτρογεννητριών και τελικά δεν μπόρεσε να ψυχρανθεί επαρκώς ο αντιδραστήρας. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Δεν πρέπει να ξαναδούμε οπωσδήποτε την αξιολόγηση κινδύνων για τα πυρηνικά εργοστάσια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να δώσει πράσινο φω για την οικοδόμηση νέων πυρηνικών εργοστάσεων σε σεισμογενεί περιοχέ, όπω η Ιταλία που έχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα ε, πυρηνικών αντιδραστήρων, ενώ είναι μια χώρα με πολλού σεισμού. Σκέφτομαι τη Βουλγαρία ή την ε, εργοστάσια όπου ε, έχουν ήδη χτιστεί πάνω σε ρήγματα και έχουν μια σχετική αξιολόγηση με παλιωμένη. Τι θα κάνει γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε και εγώ καταρχήν ε, σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ σήμερα και θέλω επίσης να πω και ένα ευχαριστώ <clears throat> για το ότι μας ε, ενημερώσετε διεξοδικά ε, για την κατάσταση ως διαμορφώνεται στην Ιαπωνία και για τα μέτρα που προτίθεστε να λάβετε. Θα πω ευχαριστώ επίσης διότι θεωρώ εσείς ως Επίτροπος αναλάβατε πλήρως την ευθύνη για αυτό αυτά που λαμβάνονται ως μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, πάρα πολύ καλό αυτό που προτείνεται τα τεστ καταπώνησης ε, των υλικών ε, και πολύ καλό που το δέχονται και τα κρατη Είναι πολύ σημαντικό να προβούμε σε νέα αξιολόγηση των κινδύνων, των προδιαγραφών. Σας παρακαλώ λοιπόν να αναζητήσετε ευρωπαϊκές λύσεις, γιατί δεν είναι δυνατόν ε, τα κράτη-μέλη μόνα τους παρά τη θέσπιση της οδηγίας του 2009. Την ξαναδιάβασα. Είναι αστείο ότι αναφέρει αυτή η οδηγία ότι δείτε ε, η ασφάλεια πρέπει να αντιμετωπίσει σε υψηλό επίπεδο. Μα δεν μπορούν αυτές να είναι οι Ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ. Κύριε Επίτροπε, σα παρακαλώ λοιπόν να ε, Υποβάλλεται νέες προτάσεις ε, και κάτι τέτοιο ε, θα τύχει και της αποδοχής ε, από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και έχω και μία ερώτηση σε σχέση με τα προτινόμενα μέτρα. Νομίζω είναι σημαντικό να σκεφτείτε το πόσο γρήγορα και καλύτερα μπορούμε να περάσουμε σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας πούμε, όσον αφορά την επέκταση των δικτύων, σκεφτήκατε μήπως ε, να επενδύσετε περισσότερα χρήματα στα έξυπνα δίκτυα. Εάν δεν ε, έχετε χρήματα θα τα ζητήσετε και ενεργειακή εξοικονόμηση ενέργειας και αποτελεσματικότητα ενέργειας. Ε, τι προβλέπετε για να επιταχύνετε τη διαδικασία. Ο συνάλφος κύριος Ρότε. Ευχαριστώ πρόεδρε και επίτροπε. Γνωρίζουμε, γνωρίζαμε όλοι ότι υπάρχει ένα ένας κίνδυνος και εμείς οι μαθηματικοί, ξέρουμε ποιος είναι αυτός, ε, αυτό είναι το υπόλοιπο κίνδυνο όπως λέγεται στα μαθηματικά, δυστυχώς το βιώσαμε την Παρασκευή. Αυτά που λέτε περί τεστ καταπονήσεως υλικών. Ε, το θέμα των ε, πυρηνικών καταλήπων αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό. Αυτά τα πυρηνικά κατάλοιπα θα συμπεριλαμβάνονται στα τεστ καταπονήσεως. Και η κυρία Χάλ το είπε πολύ σωστά. Ε, το αίτιο ε, όλης ε, αυτής της κατάστασης δεν ήταν ο σεισμός αλλά το ότι κατέρευσε η παροχή ενέργειας και προέκυψε αλυσιδωτή αντίδραση. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τα 143 πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα, πώς εξεταστούν, θα εξεταστεί ε, το έτος κατασκευής τους, ε, η διάρκεια ζωής τους, γιατί και τα εργοστάσια αυτά έχουν διάρκεια ζωής. Ε, ο παράγων αυτός και η αύξηση του υπόλοιπου κινδύνου πώς ακριβώς αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ακόμα δεν έχει γίνει σαφή αξιολόγηση των γεγονότων, ούτε ξέρουμε τι συνέβη, ούτε και τι θα συμβεί επακριβώς. Ξέρουμε όμως ότι η στάση της κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει και αλλάζει και η στάση μας προς την πυρηνική ενέργεια. Θα αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο συζητάμε την πυρηνική ενέργεια. Ήδη ακούμε ε, και το ενδεχόμενο να τροποποιήσουμε το ενεργειακό μείγμα. Θα ήθελα να σα θέσω την εξή ερώτηση, κύριε Επίτροπε. Εσεί θεωρείτε ότι τα όσα συνέβησαν στην Ιαπωνία θα πρέπει να επιδράσουν στην ενεργειακή στρατηγική που έχουμε ήδη αναλάβει. Και τι θα θέλατε να απαντήσετε εσεί σε αυτές τις χώρες που σήμερα σκοπεύουν να ξεκινήσουν την κατασκευή νέων πυρηνικών αντιδραστήρων ε, στην επικράτειά τους. Ήδη τώρα ο Πρωθυπουργό τη Βραδεμβούργου δηλώνει ότι θα πρέπει η Γερμανία να ξανασκεφτεί τα σχέδια επενδύσεων σε πυρηνική ενέργεια. Επειδή εμεί δεν έχουμε κανένα πυρηνικό ε, αντιδραστήρα και οι Γερμανοί έχουν 17. Ο κύριο Χατζημαρκά. Ε, Κύριε Επίτροπε, εσείς ε, με τα τεστ αυτά θέλετε να επιτύχετε εξευρωπαϊσμό ε, του προγράμματος αυτό. Στην Βουλγαρία Υπάρχει αντιδραστήρα. Δεν λειτουργεί, αλλά θα μπορεί να ξαναλειτουργήσει. Και το Fesselheim. Και αυτό είναι δύσκολο για τη Γερμανία. Επίσης, η Γερμανία είπε από αύριο ε, θα θέσει εκτός λειτουργία 7 πυρηνικά εργοστάσια. Αυτή η ε, πολιτική της Γερμανία μήπω σα βοηθάει στο να επιταχύνετε κι εσεί να αναζητήσετε εναλλακτικέ λύσει. <coughs> Τρίτη ερώτηση. Υπάρχουν... Ε, και άλλοι πυρηνικοί σταθμοί πάνω σε σεισμογενείς περιοχές. Δεν πρέπει λοιπόν να αξιολογήσουμε σωστά αυτούς τους ε, πυρηνικούς σταθμούς και εσείς ε, ως ε, Επίτροπος ίσως θα πρέπει να εντάξει το θέμα αυτό στις διαβουλεύσεις των, της ομάδας των G20. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ένα ερώτημα θέλω να θέσω. Μετά την προσωρινή πτώση των τιμών, πιστεύετε ότι θα ανέβει η τιμή του πετρελαίου. Η Ιαπωνία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου παγκοσμίω. Μπορούμε να, να φανταστούμε ότι θα αυξηθούν οι τιμές, θα διωγγωθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου λόγω των όσων συνέβησαν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, σκεπτόμενο στην Ιαπωνία λυπάμαι πάρα πολύ. Στενοχωριέμαι. Ε, και όταν σκέφτομαι την Ευρώπη, χάνω την υπομονή μου, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Η πτώση ενός αεροπλάνου ε, πάνω σε ένα ποινικό εργοστάσιο που δεν προστατεύεται δεν είναι πιο απίθανο από αυτά που συνέβησαν στην Ιαπωνία. Και αυτά τα δύο ε, στα μαθηματικά αποκαλούνται rest risk, υπόλοιπο κινδύνου. Αυτό λοιπόν ε, το ε, υπόλοιπο κινδύνου, γιατί δεν το αντιμετωπίζει σωστά να εξάγουμε τις απαραίτητες ε, συνέπειες και να πούμε ότι επιθυμούμε αυτόν τον κίνδυνο που μπορεί να μετρηθεί ποσοτικά, αυτόν τον κίνδυνο θα τον λάβουμε υπόψη μας. Κύριε Οτιγκέρ, πότε θα παρουσιάσετε στην κοινή γνώμη ε, τα αποτελέσματα των τεστ ε, καταπώνησης υλικών. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Επιτροπό για την ε, προθυμία του και την παρουσία του εδώ. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια των τεστ καταπονήσεως, βλέπετε ότι οι δοκιμές γίνονται σε εθελούσια βάση και διοργανώνονται από τη Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Υπάρχει μια σειρά κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη, μήπω όμω να προβλεφθούν κάποια περαιτέρω, διότι στι κάτω χώρε βλέπουμε να υπάρχουν ε, ε, κριτήρια που ισχύουν από τη δεκαετία του 70. Τα κριτήρια λοιπόν αυτά δεν πρέπει να αναθεωρηθούν και να τα συζητήσετε και μαζί μας γιατί μπορεί να αφορούν στο μέλλον ένα γεγονός που θα ελάμβανε χώρα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Ματίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, και εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Και απευθείας να θέσω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, κύριε Επίτροπε, αναφέρατε ότι ότι τα όσα συνέβησαν στην Ιαπωνία ήταν πράγματα που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν. Ας πούμε ότι συμβαίνει μια φυσική καταστροφή στην Ευρώπη. Εμείς θα μπορούσαμε να ελέγξουμε καλύτερα τα, τα όσα θα συνέβαιναν εδώ δεν θα ήταν η κατάσταση εκτός ελέγχου. Και για όσα αναφέρατε για τα τεστ καταπονήσεως και τις σχετικές προδιαγραφές, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επίπτωση αυτής της δραματικής κατάστασης που ζούμε στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την ε, πυρηνική ενέργεια. Δεν υπάρχει εδώ κάποιο μάθημα που θα πρέπει να αντλήσουμε. Επίτροπε, ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ και Έχω μία ερώτηση. Ε, αρκετοί συνάδελφοι είπαν ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε το συντομότερο δυνατόν την ποινική ενέργεια. Και εγώ θέλω αυτό να το συνδυάσω με τους στόχους ε, της προστασίας του κλίματος. Ε, μέχρι το 2020 έχουμε στόχους ε, και αυτή τη στιγμή το 32% του ενεργειακού μείγματος είναι πυρηνική ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπολογίσει μέχρι το 2020 πόσο μπορούμε να περιορίσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα χωρίς πυρηνική ενέργεια, χωρίς να χρησιμοποιούμε πυρηνική ενέργεια. Ο κύριος Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τα όσα ξεκίνησε. Οι συνέπειες ε, του ε, ατυχήματος στο Τσερνομπίλ ήταν αντίστοιχες. Ε, το σύστημα ψήξης δεν λειτουργούσε σωστά και μετά από τόσα χρόνια η Ευρώπη ακόμα δεν έχει δημιουργήσει όπως θα έπρεπε κάτι καλύτερο. Μέχρι τούδε τα πυρηνικά εργοστάσια είχαν δύο προτεραιότητες αφενός ε, ήταν προτεραιότητα ως ενέργεια γιατί ήταν η φθηνότερη και η πιο καθαρή πηγή ενέργειας. Μπορούμε να ε, επιχειρηματολογήσουμε βέβαια υπέρ του ε, θέματος της καθαρής ενέργειας, διότι έχουν νιώσει οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στο πετσί τους τους θανάτους και τα προβλήματα στην υγεία μετά από πυρηνικά ατυχήματα. Το θέμα είναι λοιπόν πόσο είναι αυτό το κόστος ε, μαζί με τη χρήση, την κατασκευή και την ρευστοποίηση των συνεπειών ε, για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτά τα τεστ καταπώνησης, αλλά είναι πολύ σημαντικό επίσης να μάθουμε όσα περισσότερα μπορούμε να μάθουμε από τα όσα συνέβησαν για να κρατήσουμε αυτά τα οποία είναι σημαντικά για, τις, για τα διάφορα ε, πυρηνικά εργοστάσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε και το γεγονός ότι η καταστροφή που συνέβη στην Ιαπωνία είναι ιστορικών διαστάσεων και, έχουν, ε, και έχει πλήξει όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Όταν κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, ε, τείνουμε να ξεχνούμε ότι καταστράφηκαν χωριά, σπίτια ε, και τμήματα πόλεων. Δηλαδή όλους τους οικονομικούς τομείς. Να φροντίσουμε όμως ότι όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από την όλη διαδικασία θα πρέπει να τα ε, δούμε και όχι μόνο μέσω των τεστ καταπώνησης αλλά να δούμε τι συνέβη και τις συνέπειές του. Μπορεί να ζούμε σε διαφορετικό περιβάλλον και να αδράξουμε όμως την ευκαιρία να βελτιώσουμε την ασφάλεια των πυρηνικών μας εργοστασίων αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ανάγκη. Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, ε, πάρα πολλές ερωτήσεις έγιναν. Όσοι δεν πήραν το λόγο θα με υβρίζουν. Τι να κάνω, θα το καταπιώ. Ε, ελπίζω κάπως καλά να τα πήγαμε, να τα μοίρασα καλά. Θέλω όμως να δώσω το λόγο στον κύριο Έτιγκερ να απαντήσει, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άλλοι 6-7 είναι. Δεν, δεν ξέρω, δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορούμε. Ναι, όλοι λένε ένα δευτερόλεπτο και εντάξει, πρέπει να φύγει ο κύριο Σότιγκερ. Θέλετε απάντηση. Είχαμε πει ποια θα είναι η διαδικασία. Ένα ε, δώσει ο κύριο Σότιγκερ ε, τι απαντήσει, γιατί μετά θα λέτε δεν έδωσε καμία απάντηση. Κύριε Ότιγκερ, σα παρακαλώ να πω το εξή ε, πριν μπούμε στην ουσία. Κοιτάξτε, εκτό συνεδριάσεων όπου καλούμεθα να απαντήσουμε, θα σας ενημερώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Και πριν αποφασίσουμε για τα τέσσερα καταπώνησης, το τι θα ελέγχθει, το ποια είναι τα κριτήρια, ε, ποιες είναι οι προδιαγραφές, ποιοι θα είναι οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και ποιοι θα επιλεγούν. Ε, πριν από κάθε απόφαση, να έρχομαι εδώ, να έχουμε χρόνο και στον διάμεσο χρονικό διάστημα να έχω επαφή με τις πολιτικές ομάδες, γιατί σήμερα είναι το εναρκτήριο λάκτισμα απλώς. Όσο δυσάρεστες και αν είναι εικόνες, διακοπή από την αίθουσα, χωρίς να ακούν οι διερμηνείς, λυπούμε πάρα πολύ, Επίτροπος. Εσείς ε, μπορείτε να με κατακεραυνώνετε, αλλά εγώ δεν θα σας πω ε, αυτά που θέλετε να ακούσετε. Προηγουμένως ήσασταν εκεί στην συνέντευξη τύπου και είπα ότι μέχρι τα μέσα του έτου ε, θα έχω ορίσει τα κριτήρια έτσι ώστε τα τεστ να γίνουν κατά το δεύτερο εξάμεινο. Μιλάει ο βουλευτής, δυστυχώς χωρίς μικρόφωνο, δυστυχώ δεν ακούν δερμηνείς και απαντάει ο Επίτροπος Αν εσείς θέλετε κύριε Τόμας να κάνετε τα τεστ, κάντε τα. Άντε και καλή τύχη. Όμως ε, στο θέμα αυτό ε, θα πρέπει να είμαστε ε, νυφάλιοι και γι' αυτό το είπα στην συνέντευξη τύπου ότι τα κριτήρια θα πρέπει να τα έχουμε διαλέξει μέχρι τον Ιούνιο, συμπεριλαμβάνοντας τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές και τις κυβερνήσεις ε, και κατά το δεύτερο εξάμεινο θα γίνουν αυτά οι δοκιμές. Είπα χωρίς καθυστέρηση, ε, αλλά ε, καλά, σωστά. Και αν γίνεται νωρίτερα, ακόμα καλύτερα. Το θέλω και εγώ. Όσον αφορά τώρα τα βασικά ερωτήματα στη σκάλα αυτή που υπάρχει, την κλίμακα μάλλον, στην κλίμακα, η Ιαπωνία κατατάσσεται στο 4. Πάλι παρατηρήσεις ε, εκτός ε, μικροφώνου. Δεν ακούμε δυστυχώς διερμηνείς. Λέω επίτροπος. Η... Συγγνώμη, γίνεται συζήτηση εκτός μικροφώνου. Πρόεδρος, ε, να κρατήσουμε κάποιους κανόνες γιατί δεν γίνεται. Και ο Επίτροπος θα πρέπει να μπορεί να τελειώσει την πρότασή του, να την πει τουλάχιστον μέχρι τέλου. Και λέει ο Επίτροπος, ίσως εσείς ε, να έχετε καλύτερη πληροφόρηση, ε, εγώ όμως θέλω να πω ότι στις 4 ώρα το απόγευμα η κατάσταση ήταν εξή. Επίσημα είναι κλίμακα 4. Οι Γάλλοι είπαν 6 και αυτή τη στιγμή δεν αποκλείω ακόμη πιο αρνητικές εξελίξεις. Επίσης, θέλω να σας πω ότι εγώ προσπαθώ να καλύψω πολλά θέματα και πέρα από τις αρμοδιότητες μου, όπως ε, πηγέ πηγές ενέργειας για το ε, ενεργειακό μείγμα μέχρι το 2020 θα είναι 33%. Στο χάρτη πορείας θα είμαστε πάνω από το 33% και αυτό θα το εξετάσουμε κατά τη διάρκεια του έτους. Δεύτερον, ανακοίνωσα την οδηγία που εγκρίνατε ε, να την αναθεωρήσουμε, να την αξιολογήσουμε νωρίτερα και να προτείνουμε νωρίτερα και ε, μία μεταρρύθμιση και περαιτέρω εμβάθυνση. Και όσον αφορά το θέμα των κρατών μελών, ε, δεν θέλω να μεταφέρω πληροφορίες από τη συνέντευξη που έλαβε χώρα προηγουμένως. Θέλω όμως να σας πω το εξή για την πυρηνική ενέργεια και για τη στάση των κρατών μελών. Εξαιρουμένου του Βερολίνου όπου ε, υπάρχει λίγη κίνηση, κατά τα άλλα δεν υπάρχει καμία απολύτως κίνηση. Η Αυστρία δεν έχει πυρηνική ενέργεια. Τι να κάνει. Παρατηρήσεις ε, εκτός μικροφώνου απάντηση του Επιτρόπου θαυμάσια. Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω για τις χώρες εκείνες που θα μπορούσαν να προβούν σε διορθώσεις στο ενεργειακό μείγμα. Αυτό αφορά την Ελβετία ως ε, γειτονική χώρα. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση ε, αφορά το δικαιοστάσιο, το μορατόριουμ, το εμπάυση λειτουργίας, ε, την εγκατάλειψη ενέργειας. Όλα αυτά όμως αφορούν τη Γερμανία. Και μπορείτε να διαμαρτύρεστε, αλλά εγώ πρέπει να σεβαστώ ε, τη στάση της γαλλικής κυβέρνησης, της Ιταλικής, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και να σεβαστώ ε, και τις τοποθετήσεις των κυβερνήσεων των νέων κρατών μελών. Γι' αυτό λοιπόν λέω να αυξηθεί το ποσοστό των νόσημων στο μείγμα, δεύτερον να εφαρμόζεται πιο αυστηρά η οδηγία, αν δείξουν τα τεστ κοπόσεως ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει πιο αυστηρή εφαρμογή. Ε, κυρία Φαν Μπρέμπτ, εσείς ε, ήσασταν χρόνια μέλος ε, κυβέρνησης της χώρας σας και αυτά τα πυρηνικά εργοστάσια ήταν εν λειτουργία όταν ήσασταν μέλος της κυβέρνησης. Δεν ξέρω εσείς τι κάνατε, αλλά για την πυρηνική ενέργεια στο Βέλγιο, εγώ μέχρι τώρα δεν έφερα ευθύνη. Εσείς Πολλά χρόνια φέρετε την ευθύνη και στην τοπική και στην εθνική κυβέρνηση. Όχι ότι θέλω να σας κατηγορήσω, μόνο που όταν ξέρουμε ότι οι εθνικές κυβερνήσεις ήταν υπεύθυνε για το ενεργειακό μείγμα και όταν εσείς ξέρετε ότι αυτά δεν άλλαξαν στη διακυβερνητική και η ε, συμφωνία ε, τήρησε αυτά τα ποσοστά, τότε ως δημοκράτες θα πρέπει να σεβαστείτε ότι τα θέματα αυτά θα πρέπει να συνεχίσουν να συζητούνται στα κόμματα και στις κυβερνήσεις. Εγώ, παραδείγματο χάρη, ε, στην Ιταλία θα γίνει δημοψήφισμα μετά από λίγες εβδομάδες για τα πυρηνικά και με Γανία περιμένω να δω το αποτέλεσμα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να κουβεντιάζετε μαζί μου, αλλά δεν θα μπορείτε να περιμένετε περισσότερα από μένα από αυτά που μπορώ να σας προσφέρω. Ο ε, Επίτροπος δεν είναι νομοθέτης, είναι εκτελεστική εξουσία και εγώ προσπαθώ να εφαρμόσω σωστά τα καθήκοντά μου και τι αρμοδιότητάς μου. Δεν μπορώ να τα υπερβώ. Αυτό είναι δική σας διακριτική ευχαίρεια και ίσως ε, μιας άλλης διακυβερνητικής με μένα μπορείτε να μιλήσετε για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς μου, αλλά για να δούμε, είμαι περίεργος να δω αν θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε περαιτέρω τη συζήτηση για το ενεργειακό μείγμα. Και θέλω να σας πω το εξής. Το φθινόπωρο, παραδείγματος χάρη, όταν θα μιλήσουμε για το 2030 και ε, το 2030 αντί να μιλάμε για 33% να πάμε πάνω από το 40% πρέπει να σας πω ότι με αγωνία περιμένω το τι θα κάνουν η Γαλλία και η Πολωνία που έχουν πυρηνική ενέργεια και άνθρακα. Κύριε Χάρμσε, αν θέλετε την επόμενη εβδομάδα να ε, συναντηθούμε, εντάξει, πολύ ωραία, μόνο που προσπαθώ τώρα, με βάση αυτά που ξέρω, να σας απαντήσω. Κάτι άλλο. Η τήξη. Όσον αφορά την τήξη του πυρήνα, αυτό μας ενδιαφέρει είναι να την αποφύγουμε. Να έχουμε σωστή ψήξη, ε, η ψήξη όμως έχει άμεση σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια. Ε, το κατά πόσον ελέγχεται η πυρηνική τήξη, αυτό πράγματι ε, και εγώ δεν το ξέρω, πολύ αμφιβάλλω. Και αν ισχύει αυτό πράγματι υπάρχουν μη αναστρέψιμες συνέπειες στο έδαφος, στο υπέδαφος. Όσον αφορά την πολιτική ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός του Τόκιο πριν από λίγες ε, ώρες ε, τοποθετήθηκε ε, στην απαράδεκτη πολιτική επικοινωνίας της επιχείρησης που λειτουργούσε αυτά τα πυρνικά εργοστάσια και τώρα απλά διαμαρτύρεται. Στην Ιαπωνία κατόπιν τούτου έχουμε μια κυβέρνηση που μπορεί να λειτουργήσει μόνο οριακά και μια επιχείρηση που λειτουργεί ταπεινικά επίση οριακή. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο όπω σα είπα. Εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέραμε κάθε μορφή τεχνική βοήθεια, αλλά τι τελευταίε ημέρε ε, διαπιστώσαμε ότι η προθυμία δεν ήταν και πολύ μεγάλη. Και μόλι πριν από λίγο απευθύνθηκαν στον Οργανισμό Ποινική Ενέργεια στη Βιέννη για να στείλει εμπειρογνώμονε. Βεβαίω το δικό μα θέμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά G20 ε, και μέσα από, την, ε, από τον Οργανισμό ε, Ποινική Ενέργειας να κάνουμε το θέμα να το φέρουμε σε διεθνέ επίπεδο. Η Ρωσία είναι εταίρο μα γιατί παίζει ρόλο στο ενεργειακό μείγμα και ίσως ε, να μπορέσουμε να εξάγουμε τα τεστ ε, καταπώνησης ε, στη Ρωσία. Ίσως το καταφέρουμε αυτό. Πράγματι, θα πρέπει όσον αφορά το ποινικό εργοστάσιο Μπελενέ στη Βουλγαρία, να ερευνήσουμε το θέμα περαιτέρω. Αυτό να το κάνει και η κυβέρνηση, να το κάνουν και οι επενδυτές. Και ας μην ξεχνάμε το εξής. Αυτή τη στιγμή η περιφερειακή αγορά χρειάζεται λιγότερες ποσότητες ενέργειας και οι επιχειρήσεις όπως οι RVS ε, αποσύρθηκαν. Κατ' ουσίαν δεν έχουν πλέον αγορά. Εκεί τουλάχιστον δεν είδα να έχουν ενδιαφέρον ε, και αποσύρθηκαν. Και τίθεται το ερώτημα κατά πόσον ε, μπορεί να εξεταστεί το θέμα της ασφάλειας. Φέστελχάιμ, το ίδιο. Και εκεί το ελληνικό εργοστάσιο Φέστελχάιμ. Πάντως, αν κάνουμε τα τεστ αυτά, θα πρέπει να παραμείνουμε αντικειμενικοί. Αυτό που έχει σημασία είναι ε, σε τελική ανάλυση το θέμα των σεισμών πρέπει να το προσέξουμε. Και τα πυρηνικά κατάλοιπα και η πυρηνική καρδιά, το σύνολο του πυρηνικού αντιδραστήριου, θα πρέπει να εξεταστεί σε αυτό να γίνει ε, τεστ καταπώνηση, αυτό είναι προφανές. Να σας πω και κάτι άλλο. Μετά το Πάσχα θα σας υποβάλουμε τα κριτήρια για τα τεστ καταπώνησης. Και με μεγάλη μου χαρά να δεχθώ τις ε, παρατηρήσεις σας πριν ε, τελικά καταλήξουμε. Και όσον αφορά τη Γερμανία, θέλω να σας πω ότι το θέμα των δικτύων, τα δίκτυα και σε διασυνοριακό επίπεδο σίγουρα θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, αυτό που παίζει ρόλο είναι και τα ορυκτά καύσιμα. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή οι αγορές ε, γνωρίζουν ε, πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Κατόπιν, θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσει το θέμα αυτό σε ανώτιτο επίπεδο, έτσι ώστε στην ομάδα G20 να στηρίξουμε τον κύριο Σαρκοζή όλοι με μια φωνή. Ε, το κατά πόσον θα αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου, αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βλέποντας τις εικόνες αυτές στην Ιαπωνία όλοι αγωνούμε ε, για τους ανθρώπους ε, και για την ενέργεια και η τιμή του πετρελαίου θα πάει 80, 90, ακόμα και 30, ε, λυπάμαι, αυτό είναι δευτερεύον. Κύριε Επίτροπε, ε, νομίζω σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων των συναντέλφων για το ότι δεν διστάσατε να έρθετε στην Επιτροπή μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναλάβατε ταχύτερα την πρωτοβουλία, ασχοληθήκατε με το θέμα αυτό και μπορείτε να είστε σίγουρος σας είμαστε ευγνώμονες για το ότι αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό με ε, ιδιαίτερα αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λύεται η συνεδρίαση.